Απευθύνω το καλό ορίσατε στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλτ Τούσκ. Έχετε το λόγο, κύριε Τούσκ. Ευχαριστώ, κύριε πρόεδρε. Κύριε πρόεδρε, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το πρόσφατο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ήταν το πιο δύσκολο τη εποχή που είμαι πρόεδρο του Συμβουλίου. Παρά το γεγονό ότι καταλήξαμε σε κοινέ λύσει, η δύσκολη καιρή είναι μπροστά μα βρίσκουμε στο Ηνωμένο Βασίλειο για το αν θα παραμείνει ή όχι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο ο λαό τη μεγάλη Βρετανία μπορεί να το αποφασίσει αυτό. Αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε από τη δική μα πλευρά, το μόνο πράγμα που μπορούσαμε να κάνουμε είναι να συμφωνήσουμε για μια νέα συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο και το πράξαμε. Τα 28 28 επικεφαλής κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκριναν ομόφωνα ένα νομοθετικά δεσμευτικό και ε, ανεπίστρεπτο σχέδιο συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο είναι σύμφωνο με τις ε, συνθήκες και δεν μπορεί να ανατραπεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Θα τεθεί όμως σε εφαρμογή μόνο αν ο Βρετανικός λαός αποφασίσει ότι η Μεγάλη Βρετανία θα μείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλιώς αυτή η συμφωνία είναι άκυρη και δεν έχει πια ύπαρξη. Συμφωνήσαμε να το κάνουμε με αυτόν τον τρόπο, ώστε να μην θίξουμε τις βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η ελευθερία διακίνησης και η αρχή της μη διάκρισης. Και χωρίς να θίξουμε τις δυνατότητες της μελλοντική οικονομικής και νομισματικής ένωσης στην Ευρώπη. Αν είχα καμία αμφιβολία για όλα αυτά, ποτέ δεν θα είχα προτείνει μια τέτοια συμφωνία. Παρά τις δυσκολίες αυτές, οι ηγέτε των κρατών τη Ευρωπαϊκής Ένωση δεν αποχώρησαν από την τράπεζα των διαπραγματεύσεων γιατί γνωρίζαμε όλοι τι διακυβεύεται. Το να κρατήσουμε το Ηνωμένο Βασίλειο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να διατηρήσουμε τη γεωπολιτική συνοχή της Ευρώπης. Θα ήθελα εδώ να εκφράσω τις ε, ειλικρινείς ευχαριστίες μου στον πρόεδρο Γιούνκερ και την ομάδα του μαζί με του οποίου εργαστήκαμε πολύ στενά σε όλη αυτή τη διαδικασία. Θα ήθελα επίση να ευχαριστήσω και του διαπραγματεύτέ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι οποίοι ήταν παρόντε σε αυτή τη διαδικασία και που ήταν πολύ αποτελεσματικοί για να μπορέσουν να επιτυχούν του στόχου που θέλαν. Πιστεύω στεναρά ότι χρειάζεται να συμμετάσχει πλήρω και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε αυτή τη διαδικασία. Πάντα θα θυμάμαι τις κέρδιες συζητήσεις με τον πρόεδρο Σούλτς, με τον ε, ηγέτη της ομάδας των φιλελευθέρων, τον κύριο Φερχόφστατ και τον Έλμαρ Μπλοκ επίσης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους μας το γεγονός ότι αυτή η συμφωνία μας επιτρέπει να λάβουμε υπόψη το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως σύνολο. Χωρίς τη βοήθειά σας αυτή η συμφωνία δεν θα ήταν εφικτή. Σας ευχαριστώ πάλι πάρα πολύ. η Ευρωπαϊκή Ένωση θα σεβαστεί την απόφαση, την ετοιμιγορία του Βρετανικού λαού. Αν η πλειοψηφία θέλει να φύγει, αυτό θα συμβεί. Αυτό θα αλλάξει για πάντα το πρόσωπο της Ευρώπης. Θα είναι μια αλλα, αλλαγή προς τα χείρο. Αυτή είναι βέβαια η προσωπική μου άποψη. Ο Πρωθυπουργό Κάμερον είπε τη Δευτέρα στη Βουλή των Κοινοτήτων ότι δεν είναι τώρα η κατάλληλη στιγμή για να διχαστεί η Δύση και δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Και αυτό έκανα ότι παίρνω από το χέρι μου για να αποτρέψω κάτι τέτοιο. Από την άλλη πλευρά, αν η Μεγάλη Βρετανία αποφασίσει να παραμείνει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ελπίζω ότι το Κοινοβούλιο αυτό θα εξασφαλίσει ότι αυτή η συμφωνία θα μεταφραστεί στην απαραίτητη νομοθεσία και θα τεθεί σε εφαρμογή αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα ήθελα τώρα να στραφώ στην κρίση μετανάστευσης. Οι ηγέτες αποφάσισαν για ένα κοινό, ότι το κοινό σχέδιο δράσης μας με την Τουρκία θα παραμείνει πρώτη προτεραιότητα και πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να μπορέσει να ευδοκιμήσει αυτό το σχέδιο. Αυτό σημαίνει σε τελική ανάλυση ότι οι μεγάλοι αριθμοί προσφύγων που βλέπουμε ακόμα να έρχονται στην Ευρώπη πρέπει να μειωθούν και αυτό να γίνει γρήγορα. Γι' αυτό έχουμε αποφασίσει να ε, διοργανώσουμε μια ειδική συνάντηση με την Τουρκία στις 7 Μαρτίου. Η συζήτηση μεταξύ των ηγετών εστίασε στο να υπάρξει μια συνένεση για την αντιμετώπιση της κρίσης. Για να το πετύχουμε αυτό πρέπει πρώτα απ' όλα να αποφύγουμε να έχουμε μια σύγκρουση μεταξύ διαφορετικών σχεδίων. Δεν έχει κανένα νόημα. Μονάχα διχασμό μπορεί να δημιουργήσει το να έχουμε σχέδιο Α, σχέδιο Β, σχέδιο Γ και αυτό δεν θα οδηγήσει σε καμία λύση. Θα πρέπει αντίθετα να προσπαθήσουμε να έχουμε μια σύνδεση, σύνθεση διαφορετικών προσεγγίσεων. Δεν υπάρχει καμία εναλλακτική λύση σε ένα πλήρες και συνολικό ευρωπαϊκό σχέδιο. Δεύτερον, η ευρωπαϊκή απάντηση δεν είναι μονάχα οι αποφάσεις που λαμβάνονται στις Βρυξέλλες. <clears throat> είναι και πολύ περισσότερο οι αποφάσεις που λαμβάνονται στις εθνικές πρωτεύουσε. Πρέπει να το αποδεχτούμε αυτό. Συγχρόνως όμως, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε το συντονισμό πίσω από αυτές τις αποφάσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται εδώ για να συνεργαζόμαστε όλοι μεταξύ μας. Και τέλος θα πρέπει να σεβαστούμε τους κανόνες και τους νόμους που όλοι έχουν συμφωνήσει και έχουμε εγκρίνει από κοινού. Αυτό αφορά τόσο τις αποφάσεις για επανεγκατάσταση όσο και την ανάγκη να επανέλθουμε σιγά σιγά σε μια κατάσταση όπου όλα τα μέλη της ζώνης του Σέγγεν εφαρμόζουν πλήρως τον κώδικα συνόρων του Σέγγεν. Δε χωρεί αμφιβολία ότι πρέπει να επαναφερθεί το Σέγγεν και θα χρειαστεί μια προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του Σέγγεν αλλά θα πρέπει να επενδύσουμε σε αυτό το σύστημα. Πρέπει να βοηθήσουμε τις χώρες αυτές να διατηρήσουν αυτόν τον κώδικα και όχι να επενδύσουμε στην κατάρρευση αυτού του συμφώνου. Το μέλλον λοιπόν του Σέγγεν θα είναι ένα από τα κέρια θέματα τα οποία θα συζητηθούν στις 7 Μαρτίου. Επίσης είναι σαφές ότι πρέπει να συνεχιστεί η ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Συρία και τους Σύριους πρόσφυγες στην περιοχή μας. Εμείς χαιρετίζουμε την σύνοδο των χορηγών στο Λονδίνο που δύο τρίτα των υποσχέσεων προήλθαν από την Ευρώπη. Οι ηγέτες αποφάσισαν να προχωρήσουν γρήγορα για την εκταμείευση των 3,3 δισεκατομμύριων ευρώ που έχουν υποσχεθεί για το 2016 και επίσης τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία αφορούν την υποστήριξη των προσφύγων στην Τουρκία. Δεν πρόκειται μονάχα για μια ευρωπαϊκή ευθύνη. Γι' αυτό εγώ θα συνεχίσω να προσπαθώ να αγωνίζομαι για μια παγκόσμια αντιμετώπιση στην κρίση αυτή στους G20 και G7 που θα συνεδριάσουν αργότερα εφέτος. Τέλος, θέλω να κλείσω με μια έκκληση να μην πάψουμε τις προσπάθειές μας. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι είμαστε ίσω την πιο επικίνδυνη στιγμή στην ευρωπαϊκή ιστορία. Θα πρέπει να δράσουμε και να έχουμε αποτελέσματα και γι' αυτό βασίζομαι στι δικέ σα προσπάθειε και υποστήριξη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Τώρα δίνω το λόγο εξ ονόματος στην Κομισιόν στον Πρόεδρο Γιούνκερ. Κύριε Πρόεδρε. Μαζί με τους Βρυτανούς φίλους κάναμε μια συζήτηση η οποία ήταν πολύ σκληρή. Η διαπραγμάτευση ήταν δύσκολη, κράτησε πολύ καιρό, αλλά μπορέσαμε, οι 27 που πήραμε μέρος και το Ηνωμένο Βασίλειο, ότι η Ευρώπη μπορεί να πάρει αποφάσεις, ακόμα και αν η κατάσταση που έχει μπροστά της είναι εξαιρετικά δύσκολη. Θέλω εδώ να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Τούσκ, ο οποίος βοηθούμενος φιλικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με κομψότητα οδήγησε στην σωστή έκβαση. Να ευχαριστήσω επίσης και τον πρόεδρο Σούλτς και τους Σέρπα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου χωρίς τους οποίους το αποτέλεσμα δεν θα ήταν αυτό το οποίο γνωρίζουμε. Καταλήξαμε σε μια συμφωνία λοιπόν με τον Βρετανό Πρωθυπουργό. Πέτυχε το μέγιστο που θα μπορούσε να πετύχει και τα κράτη-μέλη επίσης προσέφεραν τα μέγιστα που μπορούσαν να προσφέρουν. Γι' αυτό λοιπόν η συμφωνία αυτή είναι fair, είναι δίκαιη και σέβεται τις βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης λαμβάνοντας υπόψη τις ανησυχίες των μεν και τις προτάσεις των δε. Πιστεύω λοιπόν ότι ο Βρετανικός λαός, ο οποίος κατά τη διάρκεια της ιστορίας απέδειξε επανειλημμένα το θάρρος του και τη σοφία του, θα πει ναι στη συμφωνία στην οποία καταλήξαμε με την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τη στιγμή που θα εγκρίνει τη συμφωνία αυτή ο Βρετανικός λαός θα καταθέσει νομοθετικές προτάσεις στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τα κοινωνικά θέματα της συμφωνίας στην οποία καταλήξαμε. Και θα επανέλθουμε λοιπόν στα θέματα αυτά όταν οι νομοθετικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατατεθούν επίσημα. Στο τελευταίο Συμβούλιο επίσης προφανώς ασχοληθήκαμε και με το θέμα της μετανάστευσης και των προσφύγων. Δεν να υπάρχει αδράνεια για τα θέματα αυτά και ο στόχος μας είναι να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τις ε, αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και να τις εφαρμόσουμε στην πράξη για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό και επομένως θα έχουμε μια συνάντηση με τη, τους Τούρκους ομολόγους μας και με την παρουσία των 28 εκπροσώπων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μπορέσουμε να δούμε πώς θα εφαρμοστεί πλήρως η συμφωνία του, του Σέγγεν. Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μόνο με ευρωπαϊκή δράση το πρόβλημα των προσφύγων. Δεν μπορεί να υπάρξει εθνική και μόνο λύση. Μόνο εμπόδια μπορούν να δημιουργηθούν. Αυτή τη στιγμή η Κομισιόν βρίσκεται σε μια διαμάχη με την Αυστρία. Είναι μια χώρα την οποία αγαπώ πολύ, αλλά δεν πρέπει οι Αυστριακοί θεωρούν ότι μπορούν να ε, υπάρξουν δράσεις εναντίον της ε, Αυστρίας για αυτά που κάνει. Εμείς έχουμε υποστηρίξει στο παρελθόν αυτά που έχει κάνει η Αυστρία στο παρελθόν και είναι πάρα πολλά και τώρα προσπαθούμε να συμφωνήσουμε με τους ε, αυστριακούς συναδέλφους μας ότι θα μπορέσει να υπάρξει μια λύση και σε αυτό. Ο πρόεδρος Σούλτς, σας ευχαριστώ πολύ. Το λόγο λαμβάνει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, κύριος Βέμπερ. Κύριοι πρόεδροι, κύριε και κύριοι συνάδελφοι, είναι γνωστή, σα είναι γνωστή καλά η κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή. Πόλεμος από τη μια μεριά, Ουκρανία μέχρι Συρία. Έχουμε από τη μια μεριά τον Πούτιν που προωθεί έναν εθνικισμό. Έχουμε δυστυχώ χαμηλά ποσοστά ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε μια γενιά νέων ανθρώπων που ψάχνει να βρει δουλειά και όταν κανείς ατενίζει αυτήν την κατάσταση δύσκολα μπορεί να δει πως στην τελευταία συνάντηση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων το ερώτημα που τους βασάνισε είναι εάν θα ληφθούν υπόψη τα συμφέροντα του ΣΥΤΙ του Λονδίνου. Διερωτώ με εάν οι προτεραιότητε τι οποίε συζητούν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων είναι οι σωστές. Οφείλουμε να το συζητήσουμε αυτό, διότι αυτέ είναι οι επιθυμίε που εξέφρασαν οι Βρετανοί. Τα δικαιώματα του ΣΥΡΙ του Λονδίνου και τα επιδόματα που θα καταβάλλονται σε παιδιά δαπών οι οποίοι έρχονται να ζήσουν στην Μεγάλη Βρετανία. Υπήρξε αποτέλεσμα το οποίο επιθυμούμε και εμείς να στηρίξουμε. Ο Ντέιβιτ Κάμερον αγωνίστηκε και πέτυχε ένα στέρεο πόρισμα υπέρ του Βρετανικού λαού. Ένα στέρεο αποτέλεσμα. Εμείς διαπιστώνουμε ότι εάν τελικώς οι Βρετανοί αποφασίσουν υπέρ της παραμονής της χώρας τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θα παίξει έντιμα τον ρόλο του για την εφαρμογή της συμφωνίας αυτής. Τρίτη διαπίστωσή μου, το αποτέλεσμα οφείλει να γίνει σεβαστό. Αυτοί που βγαίνουν τώρα στη Μεγάλη Βρετανία και λένε ότι εάν ο κόσμος πει όχι θα υπάρξει και άλλη διαπραγμάτευση και επομένως ενδέχεται το αποτέλεσμα να γίνει ακόμα καλύτερο, νομίζω ότι δεν υπηρετούν την αλήθεια. Τουλάχιστον για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα δεν θα υπάρξει παραπέρα διαπραγμάτευση. Κυρίε και κύριοι, οι Βρετανοί προχωρούν τώρα στη συζήτηση και αυτοί τελικώ θα αποφασίσουν. Πρώτα-πρώτα φοβάμαι ότι θα ταλαιπωρηθεί η αλήθεια. Άκουσα τον Νάιζελ Φάραντζ να λέει ότι οι εμπορικές σχέσεις είναι πολύ καλύτερες και ευκολότερες για την Μεγάλη Βρετανία εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διορωτώ με γιατί το μεγαλύτερο εμπόριο το έχει η, Ευρωπαϊ... το έχει η Ομοσπονδική Γερμανία η οποία είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί η Ιρλανδία, γιατί παρακαλούν οι Αμερικανοί και οι Κινέζοι τη Μεγάλη Βρετανία να παραμείνει εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Νάτζελ Φάρατζ ισχυρίζεται ότι 5.000 αλλοδαποί μαχητές πηγαίνουν προς την, Μεγάλη Βρετανία. Βεβαίως αυτά τα γνωρίζει μόνο διότι η χώρα του συμμετέχει στην Ευρωπόλ. Τι θα γίνει όταν θα φύγει από αυτό. Ο Νάντζελ Φάραντς λέει πολλές αναλήθειες για να παραπλανήσει τους Βρετανούς ψηφοφόρους. Το άλλο ερώτημα είναι ποιος θα χάρει εν τέλει εάν ψηφίσουν αρνητικά οι ε, Βρετανοί. Ο Πούτιν και οι τρομοκράτε θα χαρούν, διότι θα τρίβουν τα χέρια του, θα μπορούν να κάνουν πολύ καλύτερα και ευκολότερα τη δουλειά του. Τρίτο, εμεί το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να απευθύνουμε πρόσκληση. Να το παλέψουμε όλοι μαζί. Ζούμε σε μια εποχή μεγάλων αβεβαιοτήτων. Αυτό πρέπει να το δει ο κάθε ένας αντικειμενικά. Μια Ευρώπη διχασμένη είναι ασφαλώς πιο αδύναμη να αρθεί στο ύψος των προκλήσεων. Γι' αυτό η πρόσκλησή μου προς του Βρετανούς ψηφοφόρους είναι να παραμείνουν κοντά μας. Λίγα λόγια για το μεταναστευτικό. Τι να πω εδώ. Σωστά τα περιέγραψε ο ε, πρόεδρος της Κομισιόν ότι επιβεβαιώθηκαν τα ήδη συμφωνημένα. Ωραίο είναι αυτό. Καλό είναι αυτό. Από την άλλη μεριά δυστυχώς βλέπω να ξεπηδούν πολλοί εθνικοί εγωισμοί και πολλοί κομματικοί εγωισμοί και δυστυχώς από όλα τα κόμματα, το σημειώνω αυτό. Αν θέλαμε να το δούμε θετικά, θα έλεγα ότι το commitment, η δέσμευση, είναι ξεκάθαρη ότι οφείλουμε να στηρίξουμε και την πρωτοβουλία του ΝΑΤΟ για την φύλαξη των εξωτερικών συνόρων και στο Αιγαίο. Και είναι σημαντικό. Οι άνθρωποι τώρα που εγκαταλείπουν το, το Χαλέπι, επειδή τους βομβαρδίζουν οι Ρώσοι, δεν μπορούμε να τους αφήσουμε στη μοίρα τους έξω από τα τουρκικά σύνορα. Δεν μπορούμε όμως να παρακαλούμε την Τουρκία να ανοίξει τα σύνορά της προς το Θαλέπι από την άλλη μεριά να κλείσει τα σύνορά της προς την Ελλάδα. Είναι και αυτό μια αντίφαση που είναι πάρα πολύ δύσκολο να λυθεί. Έτσι λοιπόν τα δύο αυτά πράγματα πρέπει να είναι ταυτόχρονα, δηλαδή και άνοιγμα των σύνορων αλλά και προσφορά βοήθειας. Όμως λόγια είπαμε πολλά. Η ώρα ήρθε να προχωρήσουμε σε έργα. Το Ίδρυμα Μπέρτελσμαν προ λίγων ημερών εξέδωσε αντιπροσωπευτική μελέτη σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχοντας ρωτήσει πολίτες απλούς. Και εκεί αυτοί μας αναθέτουν δύο καθήκοντα. Αφενός, 79% των Ευρωπαίων θέλουν να διατηρηθεί η ελευθερία διακίνησης μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και 60% των Βρετανών, σημειώστε, επιθυμούν να παραμείνει η ελεύθερη διακίνηση. Και 67% των Ευρωπαίων θέλουν να βοηθήσουμε τους πρόσφυγες. Και αυτό όλοι μαζί οι πολίτες της Ευρώπης εμφανίζονται πολύ ευφιέστεροι από ό,τι καμιά φορά η πολιτική τους. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Κάρβερ, θέλω να σας θέσει ένα ερώτημα. Κύριε Κάρβερ, έχετε. Ο κύριος Κάρβερ, λοιπόν. Ευχαριστώ κύριε βέβαια. Θέλω να επαναλάβετε αυτό που είπατε. Είπατε ότι η επαναδιαπραγμάτευση είναι η τελική επαναδιαπραγμάτευση. Γιατί ορισμένοι δίνουν την εντύπωση του Βρετανούς εκλογή ότι θα υπάρξει ένα δημοψήφισμα και μετά θα επανέλθουμε και θα ξαναρχίσουμε τις διαπραγματεύσεις. Για λόγους σαφήνες μπορείτε να διαβεβαιώσετε το λαό του Ηνωμένου Βασιλείου ότι είναι η τελευταία διαπραγμάτευση και θα υπάρξει περαιτέρω αναδιαπραγμάτευση μετά από το δημοψήφισμα. Ευχαριστώ. Ο πρόεδρος Βέμπερ, αν χρειάζεστε διευκρίνηση των όσων ήδη είπα, ευχαρίστω να σας την δώσω. Η πρόταση έχει κατατεθεί. Πρόκειται για μια προσφορά και προς τις δύο πλευρές. Συμβιβασμό αυτό σημαίνει ότι και οι δύο πλευρέ κινούνται η μια προ την άλλη. Αυτό είναι η ιδέα του συμβιβασμού και οι δύο πλευρές κατέβαλαν προσπάθειες. Έχει λοιπόν γίνει η πρόταση, ελπίζουμε ότι η Βιτ Κάμερον και όλοι όσοι είναι υπέρ ενός κοινού μέλλοντος θα μπορέσουν να πείσουν τον Βρετανικό λαό. Αν όμως βγει το, ναι, το, συγγνώμη, το όχι από το δημοψήφισμα δεν θα υπάρξει άλλη αναδιαπραγμάτευση. Ευχαριστώ, λέει ο Το λόγο λαμβάνει ο κύριος Πιτέλα εξ ονόματος Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Θα ήθελα να διευκρινίσω εξ ονόματος της πολιτικής μου ομάδας το εξή. Το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι γιατί αυτό θα ήταν απλά βολικό. Όλοι γνωρίζουμε ότι ένα πιθανό Brexit θα ήταν ένα άλμα στο κενό, με καταστροφικές συνέπειες, ιδιαίτερα για τους ίδιους τους Βρετανούς. Όμως η Ευρώπη με το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχει παντρευτεί από συνοικέσιο. Είναι τμήμα της Ευρώπης το Ηνωμένο Βασίλειο και εμείς λοιπόν όπως και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε μια κοινή ιστορία, ένα κοινό πολιτισμό και χωρίς το Λονδίνο, χωρίς το Ηνωμένο Βασίλειο η Ευρώπη θα ήταν διαφορετική. Άκουσα για τη συμφωνία της Παρασκευής, θέλω να ευχαριστήσω όλους πήραν μέρος και τον κύριο Σούλτς και του Σέρπα και την Επιτροπή και τους φίλους του Συμβουλίου για την προσπάθεια που έκαναν. Θέλω όμως να προσθέσω το εξής, ότι εμείς δεν θα δεχθούμε να γίνουμε όμοιροι κάποιων εσωτερικών ισορροπιών του Βρετανικού Συντηρητικού Κόμματος. Είναι απαράδεκτο γιατί αυτή τη στιγμή η Ευρώπη υφίσταται τη χειρότερη κρίση της ιστορίας της. Αλλά συζητάμε στο Συμβούλιο για τη στάθμιση των ψήφων ή τι θα γίνει ακριβώς με την Τραπαζική Ένωση. Η Συμφωνία της Παρασκευής λέει ότι σε νομικό επίπεδο η αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών δεν φύγεται. Το σημειώνω αυτό θετικό αλλά όμως υπάρχει κάτι το οποίο δεν με πείθει, είναι το κοινωνικό κομμάτι. Ας φανταστείτε δύο νέους ανθρώπους, δύο Ευρωπαίους νέους που κάνουν την ίδια δουλειά. Κινδυνεύουμε με τη νέα ρύθμιση ένας από τους δύο, επειδή δεν είναι Βρετανός, έχει λιγότερα δικαιώματα από τον άλλο. Αυτό είναι διάκριση. Αν και ελπίζω, εκφράζω την ελπίδα, ότι θα διαψευστώ από τις προτάσεις τις οποίες θα παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά την έκβαση του Βρετανικού Δημοψηφίσματος. Υπάρχουν για μας κάποιες βασικές αρχές, κόκκινες γραμμές, τις οποίες πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί, γιατί αλλιώς μπορεί να κάνουμε πράγματα ανεπανόρθωτα. Δεν πρέπει να υπάρξουν διακρίσεις για τους πολίτες της Ένωσης θα δώσουμε μάχη για να παραμείνει το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το λέω αυτό, σεβόμενος τους Βρετανούς πολίτες και αυτοί φυσικά είναι κυρίαρχοι, μόνον αυτοί ε, θα αποφασίσουν και το λέγω αυτό με κάθε σεβασμό. Εσείς έχετε σταθεί πρωταγωνιστές παγκόσμιοι, ήσασταν υπέρ της ειρήνης, ήσασταν υπέρ της δημοκρατίας. Αυτές ε, οι αξίες χαρακτηρίζουν το DNA του Ηνωμένου Βασιλείου. Λοιπόν, πού αλλού θα αποδείξετε καλύτερα αυτές τις αρχές παρά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα ξεπεράσουμε τις προκλήσεις ε, θα ξεπεράσουμε τους φόβους, θα αντιμετωπίσουμε την υψηλή ταχύτητα της παγκοσμιοποίησης, γιατί το να μένει κανείς μόνος η μοναξιά είναι θλίψη, είναι εγκατάλειψη, ενώ αν είμαστε μαζί θα είμαστε δυνατοί. Ευχαριστώ κύριε Πιτέλα. Ο κύριος Πάτιν θέλει να σας θέσει μια ερώτηση αν επιτρέπετε. Thank you very much, Mr. President. Thank you, Mr. Um, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και σας κύριε Πιτέλα. Παρακαλώ μια διευκρίνηση. Αν κατάλαβα καλά το νόημα των λόγων σας, φαίνεται να εννοείται ότι δεν θα υπάρχει διάκριση στα κοινωνικά δικαιώματα όπως και αν έχει η συμφωνία του κ. Κάμερον, λέει πάντως ότι για ένα διάστημα θα καταβάλουμε επιδόματα παιδιών στο ύψος αυτών που ισχύουν στην χώρα της προέλευσής τους και όχι αυτό, στο ύψος του, ε, του Ηνωμένου Βασιλείου. Θα δούμε τι θα γίνει όταν η νομοθεσία αυτή θα έλθει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όμως λέτε ότι η νομοθεσία που θα έλθει εδώ θα είναι διαφορετική από, την, ε, από το περιεχόμενο της συμφωνίας. Τι λέτε ακριβώς δηλαδή ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να τροποποιήσει την ε, ρύθμιση που προβλέπει η συμφωνία. Κοιτάξτε, είστε ευρωβουλευτής, γνωρίζετε όπως και εγώ, πρέπει τουλάχιστον να γνωρίζετε τις διαδικασίες. Εγώ δεν προσπαθώ να εφεύρω τίποτα. Εμείς εκφράζουμε την ευχή ότι οι Βρετανοί θα υπεψηφίσουν την πρόταση και θα παραμείνει το Ηνωμένο Βασίλειο και μετά από αυτή τη σημαντική στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να καταθέσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που είναι συνομοθέτης τα εφαρμοστικά μέτρα και τότε θα γίνει ξανά μια συζήτηση. Κανένα κοινοβούλιο ελεύθερο και αυτόνομο δεν μπορεί να προβλέψει το αποτέλεσμα πάνω σε κάτι το οποίο δεν γνωρίζει. Όταν θα προταθούν τα μέτρα εμείς θα τα εξετάσουμε με επικοδομητικό πνεύμα, γιατί εμείς όπως και να έχουν τα πράγματα θέλουμε να παραμείνετε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ευχαριστώ κύριε Πιτέλα. Ο κύριος Φόξ, εξ ονόματος της ομάδας ε, Ευρωπαίων Δημοκρατών και Μεταρρυθμιστών. Thank you, President. The deal struck last week. Η συμφωνία στην οποία καταλήξαμε την προηγούμενη εβδομάδα ήταν μια σκληρή συμφωνία. Πολλές χώρες είχαν ανησυχίες, είχαν αντιρρήσεις, αλλά μπορέσαμε να τις ξεπεράσουμε. Βοηθηθήκαμε από την ισχυρή θέληση, με αντοχή ε, μπορέσαμε να βρούμε μια πρόταση. Καταλήξαμε σε μια συμφωνία η οποία καθιερώνει ένα ειδικό καθεστώς για το Ηνωμένο Βασίλειο που ποτέ δεν ήταν και δεν θα είναι στο ευρώ, στην ευρωζώνη ή στο Σέγγεν. Δεν θέλουμε να είμαστε τμήμα μιας πολιτικής διαδικασίας η οποία οδηγεί σε συμφωνίες αμφίβολες ε, ε, σύμφωνα με την άποψή μας. Εμείς θα συνεχίσουμε να παίζουμε το ρόλο μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να υπάρχουν διακρίσεις. Η ομάδα των Βρετανών συντηρητικών λοιπόν λέγει ότι η κατάληξη αυτή ήταν θετική και θα πρέπει να κρίνει ο Βρετανός εκλογέας. Εγώ θα υποστηρίξω την εκστρασία να παραμείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Easy, gentlemen. Ηρεμία. Το λόγος για τον οποίο το κάνω αυτό είναι εξή. Η ανάκαμψη οικονομική της Μεγάλης Βρετανίας είναι καλή μεν, αλλά είναι εύθραυστη και δεν θα ήθελα να τη θέσουμε σε κίνδυνο φεύγοντας από την ενιαία αγορά. Νομίζω ότι οι εκλογή μου θα είναι ασφαλέστερη, η χώρα μου θα είναι ασφαλέστερη αν μπορέσουμε να συνεργαζόμαστε πάντα με τους Ευρωπαίους εταίρους. Είναι καλοί βέβαια άνθρωποι αυτοί που διαφωνούν μαζί μου και σέβομαι τις αποφάσεις τους. Αν ο Βρετανικός λαός αποφασίσει να φύγουμε τότε θα εφαρμόσουμε την επιλογή αυτή. Υπάρχουν όμως και κάποιοι οι οποίοι δεν σέβονται τις αποφάσεις των άλλων και τις απόψεις των άλλων. Αυτοί που φωνασκούν, αυτοί που συγκρίνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Σοβιετική Ένωση. Είναι παράλογο, ανόητο και προσβλητικό για αυτούς που έζησαν κάτω από τον κομμουνιστικό ζυγό. Because unlike Αντίθετα με την Σοβιετική Ένωση, κάθε χώρα μέλος είναι ελεύθερη να φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι λοιπόν η άποψη του κυρίαρχου λαού. Το να είμαστε στην Ένωση είναι μια επιλογή και εμείς σαν κόμμα σεβόμαστε την επιλογή αυτή. Οι ψηφοφόροι λοιπόν στο Ηνωμένο Βασίλειο θα ασκήσουν το δικαίωμά τους αυτό. Θα αποφασίσουν αυτοί αν θα μείνουν ή αν θα φύγουν και στο Ηνωμένο Βασίλειο μπορούμε λοιπόν εμείς τους επόμενους τέσσερις μήνες θα συζητήσουμε ακριβώς το θέμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αντιμετωπίσει τη μεταναστευτική κρίση βέβαια. Ο Ολλανδός Πρωθυπουργό είπε ότι έχουμε 6 με 8 εβδομάδες για να σώσουμε το Σέγγεν. Το είπε αυτό εδώ και πέντε εβδομάδες. Σε αυτό εδώ το σώμα βλέπουμε κάποιους που δέχονται ότι η μεταναστευτική κρίση ε, πραγματικά οξύνθηκε όταν η, Αγγέλο, η Αγγέλα Μέρκελ είπε ότι θα δεχθεί τους ανθρώπους χωρίς όρια και θα τροποποιηθούν οι κανόνες ε, και βέβαια έρχονται οι άνθρωποι αυτοί χωρίς ανώτατα αριθμητικά όρια. Κάποιες χώρες όπως η Ουγγαρία υπερασπίζονται τα σύνορα, εφαρμόζουν τους κανόνες και τους υφίσταται κριτική, ενώ άλλες χώρες που παραβιάζουν τους κανόνες χειροκροτούνται. Δεν μπορούμε εμείς να ξεκινήσουμε να λύνουμε την κρίση αυτή αν δεν εφαρμόσουμε τους ισχύοντες κανόνες. Πρέπει να προστατεύσουμε τα εξωτερικά σύνορα. Πρέπει να βοηθήσουμε να χαμηλώσουμε τις εντάσεις τις μεταναστευτικές, να διευκολύνουμε τις επιστροφές, τις επαναπροωθήσεις απαιτείται να υπάρξει διεθνής δράση για να τελειώσει η σύγκρουση στη Συρία. Πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στους πρόσφυγες που είναι ήδη σε στρατόπεδα στο Λίβανο, την Ιορδανία και την Τουρκία. Πρέπει να τους βοηθήσουμε και με καταφύγιο δίδοντάς τους αλλά και ανθρωπιστική βοήθεια. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει προτεραιότητα σε αυτούς που διασχίζουν το Αιγαίο ή μήπως αυτούς που ήδη είναι ταξινομημένοι από τα Ηνωμένα Έθνη. Κύριε Τάσκα, στην επόμενη συνάντηση κορυφής θα πρέπει εσείς να πείτε στους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι έχουν καθυστερήσει. Σας ευχαριστώ κύριε Φόξ. Ε, υπάρχει ερώτηση του ε, βουλευτού κύριου Κόρμπετ, αν δέχεστε. Ρίτσαρτ Κόλβετ. Με χαρά άκουσα τον κύριο Φόξ να λέει ότι τάσεται επιτέλους υπέρ της εκστρατείας να παραμείνει η Βρετανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γνωρίζουμε ότι είναι διχασμένη η χώρα στο ερώτημα αυτό. Ρωτώ, μεταξύ των 20 Βρετανών συντηρητικών ευρωβουλευτών πόσοι έξιμών θα συμπαραταχθούν με τον Πρωθυπουργό σας υπέρ της παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πόσοι θα συμπαραταχθούν με το κόμμα UKIP για να αποχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση χτυπώντας δυνατά την πόρτα. Ορίστε κύριε Φόξ. Κύριε Πρόεδρε, εφόσον ενδιαφέρεται τόσο πολύ για τις απόψεις των συναδέλφων μου και ο Σκόρμπετ, ας έρθει να τους ρωτήσει προσωπικά. Φιλελεύθερη ομάδα, ο κύριος Βερχόφστατ. Παρ' όλα αυτά μου φάνηκε ενδιαφέρουσα η ερώτηση του κύριου Κόρμπετ και νομίζω ότι μπορώ να συμπληρώσω. Η κυρία Γκουλά... είναι, είναι σίγουρα διαδικαστικό το θέμα, η κυρία Γκουλάρ. Ναι κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι είμαστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όταν δίδετε τις μπλε κάρτες θα πρέπει να βλέπετε και μένα, θα πρέπει να διευκολύνετε τις συζητήσεις ανάμεσα στους Βρετανούς και άλλους εκπροσώπους και όχι να κάνετε μία συζήτηση μεταξύ των Βρετανών που μπορεί να γίνει σε άλλους χώρους. Γι' αυτό ακριβώς θα ήθελα να ζητήσω εκ νέου τη δυνατότητα να θέσω ένα ερώτημα προς τον κύριο Φόξ. Ο πρόεδρος Αγαπητή ο κανόνας που ισχύει στο σώμα είναι ότι η γαλάζια κάρτα προηγείται λόγω ταχύτητας και όχι λόγω εθνικότητας. Ο κ. Κόρμπερτ ήταν ταχύτερος. Δίνω κάθε φορά στην πρώτη γαλάζια κάρτα. Εκτός από τον κ. Μπέλεν Κέναμιν που είχε ζητήσει το λόγο ήδη πριν να λάβει το λόγο ο συνάδελφος τοποθετήθηκε. Βεβαίω ισχύει αυτό. Πώ μπορείτε να ισχυρίζετε κάτι τέτοιο, κυρία συνάδελφε. Δεν έχει μικρόφωνο η κυρία συνάδελφος. από εδώ εγώ βλέπω τουλάχιστον το ίδιο καλά όπως εσείς και είναι σαφέστατο για μένα ότι ο κ. Κόρπετ ζήτησε πρώτο τη γαλάζια κάρτα. Αν είχατε ζητήσει πρώτη εσεί, θα είχατε λάβει εσεί τον λόγο. Τώρα θα μιλήσει ο πρόεδρο τη δική σα κυρία, ε, κυρία Γκουλάρ πολιτική ομάδα, ο κ. Βεχόστατ. Για να συνεχίσω στο ερώτημα του κυρίου Κόρπετ και τη κυρία Γκουλάρ. Αναρωτιέμαι κύριε Φόξ, γιατί μιλάτε εσεί και όχι ο κύριο Καμάλ φαίνεται ότι δεν ξέρετε ακόμα τι θα κάνετε. Και αυτό ίσως είναι μια πιο εύγλωτη απάντηση στο ερώτημα του κυρίου Κόρμπετ παρά να του πείτε να ρωτήσει τους βουλευτές της ομάδας. Έχω ένα άλλο ερώτημα. Εγώ ήμουνα στη διαπραγματεύση από την αρχή, κύριε Φόξ. Και πάντα αναρωτιόμουν γιατί η Μεγάλη Βρετανία είναι τόσο ζωτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η συμφωνία γιατί είναι τόσο ζωτική. Να σας πω ότι αυτή είναι μια συμφωνία όχι για την Ευρώπη, αλλά μια συμφωνία επανένωσης μέσα στο κόμμα των Τόριδων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν ξέρω ποιο είναι το αποτέλεσμα βέβαια του δημοψηφίσματος, αλλά ένα αποτέλεσμα είναι σίγουρο για μένα. Δεν θα επανενωθεί το κόμμα των συντηρητικών, η Τόρις, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Γιατί βλέπω όλο αψιμαχίες μεταξύ σας για το θέμα αυτό. Ο Τζόνσον να προκαλεί τον Ντέβιτ Κάμερον και εγώ είμαι φιλόδοξος πολιτικός και καταλαβαίνω τον Μπόρις Τζόνσον. Αλλά ίσως το φέρνει σε άλλο επίπεδο ο Μπόρις και τον παρατραβάει λιγάκι. Γιατί έχουμε τον ε, δήμαρχο του Λονδίνου να δρά εναντίον του πρωθυπουργού της χώρας τους. Δεν ξέρω λοιπόν αν αυτό είναι μια φιλοδοξία για καλύτερη Μεγάλη Βρετανία και μια καλύτερη Ευρώπη είναι νομίζω κάτι το οποίο είναι λυπηρό, δεν έχει νόημα. Είναι και ακόμα και για την Μεγάλη Βρετανία κάτι δραματικό. Βλέπουμε λοιπόν να χάνεται αυτό το οποιαδήποτε έννοια ενότητος και σταθερότητος και έχουμε τους ε, Αμερικανού να χρειάζεται να παρεύουν και να πούν δεν θα κάνουμε καμία συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο εκτό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάει και η ειδική σχέση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ηνωμένου Βασιλείου. Δεν είναι πια τόσο ειδική αυτή η σχέση. Θα σα δώσω λοιπόν κάποια συμβουλή σε αυτού οι οποίοι κάνουν αυτή τη συζήτηση μέσα στη Μεγάλη Βρετανία. Τον μη θεωρήσετε ότι μετά από ένα όχι θα μπορέσετε να γυρίσετε στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων. Γιατί αυτό το έχουν κάποιοι στο μυαλό του. Λέγοντα Α, Ευρώπη είναι. Λέτε ναι, λέτε όχι σε ένα δημοψήφισμα, σου λένε ελάτε να τα ξαναβρούμε. Όπως έκανε η Δανία, όπως έκανε η Γαλλία και οι κάτω χώρε. Αλλά εδώ δεν έχουμε το ίδιο πράγμα. Αυτό αφορούσε το Σύνταγμα της Ευρώπη. αυτό αφορούσε μια συνθήκη. Εδώ είναι ή είσαστε μέσα ή είσαστε έξω. Ή το ένα ή το άλλο. Και αν δω πώς πήγε προ τα κάτω βουτιά η Βρετανική Λύρα. Πώς βλέπω ότι έχει αποξερωθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες η Μεγάλη Βρετανία και πώς σιγά σιγά το Ηνωμένο Βασίλειο γίνεται η μικρά Αγγλία, τότε η δική μου συμβουλή θα ήταν να παραμείνετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά αγαπητοί συνάδελφοι, αυτή η συζήτηση μπορεί να έχει ένα θλιβερό χαρακτήρα, αλλά παρόλα αυτά είναι μια σημαντική συζήτηση για την Ευρώπη. Αυτό το οποίο συζητάμε σήμερα μας τονίζει ότι είναι απαραίτητη η ενότητα και όχι ο διχασμός. Ποιοι κερδίζουμε από μία Ευρώπη που είναι διχασμένη. Άνθρωποι σαν τον Βλαντιμίρ Πούτιν, τον Μπασάρα Λασάντ, το Ισλαμικό κράτος. Επομένως, αντί να σκεφτόμαστε πώς θα αντιμετωπίσουμε από κοινού όλους αυτούς, να έχουμε μια κοινή στρατηγική, δείχνουμε διχασμό, διαιρέσεις, αδυναμία και χθε έγινε πάλι σαφές όταν το Αμερικανοριστικό σχέδιο για την κατάπαυση του πυρός στη Συρία έγινε απουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ληφθεί μια σημαντική απόφαση. Μπορούμε να συνεχίσουμε. Και κάποιοι το συνεχίζουν. Μπορούμε να συνεχίσουμε να, διαπρα... διαμαρτυρόμαστε για αυτή τη συμφωνία και για τις αρνητικές της πτυχές. Η δική μου έκκληση κύριε Πρόεδρε και κύριε Τάσκ και σε όλους εδώ κάντε το αντίθετο. Ας χρησιμοποιήσουμε αυτή τη συμφωνία για να ξαναγυρίσει η Ευρώπη στις ράγες, για να μπορέσει και πάλι η Ευρώπη να λειτουργήσει. Ας σταματήσουμε την Ευρώπη à la carte. Ας σταματήσουμε την αδράνεια που οφείλεται στο βρετανικό θέμα. Δεν έχω τίποτα κύριε Φόξ εναντίον του να έχει ειδικό καθεστώ η Μεγάλη Βρετανία. Εάν την επόμενη φορά συμφωνήσετε επίση ότι την επόμενη φορά που θα γίνει μεταρρύθμιση της ε, συνθήκη θα υπάρξει και μία μεγαλύτερη ολοκλήρωση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί το χρειαζόμαστε να αντιμετωπίσουμε τι πολλαπλέ κρίσει που έχουμε ενώπιόν μα σήμερα και προφανώ την κρίση των προσφύγων. Και αυτή είναι η τελευταία μου παρατήρηση. Πρέπει να κάνουμε περισσότερα για την κρίση των προσφύγων. Να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να λύσουμε, κύριε Τόσκ, το πρόβλημα αυτό, τουλάχιστον τι ίδιε προσπάθειε που έγιναν για να λυθεί το θέμα του Brexit. Ευχαριστώ. So, Εφτά συνάδελφοι θέλουν να σας θέσουν ερωτήσεις. Εφτά. Απάντηση χωρίς μικρόφωνο. Η... Όμως η αγανακτή σας συνάδελφό συνάδελφός σας έχει ήδη αποχωρήσει από την αίθουσα. Έχω 7 λοιπόν. Η πρώτη συνάδελφος που ζήτησε όσο το λόγο είναι η κυρία Γιάκον Σάρη από την Φιλανδία, φανταστείτε. μια φιλανδή συνάδελφο επιθυμεί να θέσει ερώτηση στον Βέλγο πρόεδρο της πολιτικής ομάδας των φιλελευθέρων. Σας ευχαριστώ κύριε πρόεδρε, ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο, ευχαριστώ και εσάς κύριε Φερχόφστατ που δέχεστε να απαντήσετε. Έχω να σας πω το εξή. Εγώ είμαι ενθουσιώδης Ευρωπαία και θέλω να σας δώσω ένα ξεκάθαρο ερώτημα. Γνωρίζετε ότι ορισμένες χώρες μέλη α, υπάρχουν και εκεί δυνάμεις που είναι υπέρ της εξόδου της Βρετανίας. Εγώ δεν βλέπω απολύτως κανένα ενδιαφέρον σε κάποιο Φιλανδό να τάσεται υπέρ της Βρετανικής εξόδου. Οι Βρετανοί θα αποφασίσουν, οι Βρετανοί ψηφοφόροι και θα τοποθετηθούν οι Βρετανοί πολιτικοί. Εάν υπάρχει πάντως ένα κόμμα στο Ενωμένο Βασίλειο που θα αγωνιστεί υπέρ της παραμονής, σίγουρα είναι το φιλελεύθερο δημοκρατικό κόμμα αυτό. Αυτά λοιπόν η κυρία Τσίμερ της ε, ομάδας της Ενωτικής Αριστεράς. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, αποτέλεσμα ενδοκομματικών διαφορών κύριε Πρόεδρε, όπου κινδυνεύει τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση να χάσει ένα σημαντικό στήλο που είναι αυτός της κοινωνικής συνοχής. Τι θα γίνει τότε με το τριπλό α, κύριε Πρόεδρε της Κομισιόν, με το τριπλό α της αξιοπιστίας. Όλες οι αποσχέσεις καταραίουν. Θα σας πω και το εξή. Πορευόμαστε προς ένα ακραίο φιλελεύθερο μοντέλο των Βρετανών. Μπορείτε λοιπόν να πείτε ότι αναζωογονήθηκε το πνεύμα της Μάργαρετ Τάτσερ στις 4 Φεβρουαρίου 2016. Το αληθινό δράμα παίζει αλλού όμως και σήμερα ακόμα. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι έφτασαν στην Ελλάδα τους τελευταίους μήνες και η άρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να τηρήσει τις δεσμεύσεις ανακατανομής των προσφύγων αυτών, διαμοιρασμού των προσφύγων αυτών. Ενώ υπάρχουν αποφάσεις, τις οποίες όμως δεν επικρίνατε εσείς, το ότι ήρθεσαν οι υποσχέσεις αυτές μόλις δόθηκαν. Μία μέρα μετά από την διάσκεψη κορυφής ανατράφηκαν οι αποφάσεις αυτές. Ενώ είχατε υποσχεθεί ότι θα μείνουν μέχρι αρχές Μαρτίου ανοιχτά τα σύνορα. Τώρα διεξάγεται στη Βιέννη διάσκεψη Βγάζοντα απ' έξω την Ελλάδα που είναι ο βασικός παίχτη στην υπόθεση αυτή. Πώς θα καταλήξουμε σε ευρωπαϊκή λύση, ούτε ακούω καμιά επίκριση για τις πρακτικές αυτές τη Βιέννης, ούτε από το Συμβούλιο, ούτε από την Κομισιόν. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι, επιτέλους, το είπατε και εσεί ο ίδιο, κύριε Γιούνκερ, να τηρήσουμε τα υπεσχημένα. Αυτή είναι και η πρώτη προϋπόθεση, ώστε να δεχθεί η κάθε χώρα τους, τον αριθμό προσφύγων που έχει υποσχεθεί ότι θα δεχτεί. Εδώ χρειάζεται συγκεκριμένη βοήθεια προς την Ελλάδα. Δεν μπορούμε να κάνουμε σαν δήθεν τα αφήνουμε αυτά σε κάποιες χώρες μέλη. Οι χώρες μέλη έχουν καθήκον να τηρήσουν τα υπεσχημένα, να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους. Αυτό είναι η ύψιστη ανθρωπιστική αξία. Και θα πω το εξή, πολύ συγκεκριμένο. Δώστε παράδειγμα. Ας λάβουν το παράδειγμα της νέας πορτογαλικής κυβέρνησης η πρόσφορα του Κώστα προς τον Τσίπρα να δεχτεί στην Πορτογαλία χιλιάδες πρόσφυγες ή πάρτε την ισπανική περιφέρεια της Βαλένθια που έχει υποσχεθεί ότι θα δεχτεί ασθενείς πρόσφυγες για να τους περιθάλψει από το Αιγαίο. Αυτά είναι τα παραδείγματα και όχι ένα παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα στον Μπόρις Τζόνσον και στον Ντέιβιτ Κάμερον που δεν με αγγίζει σε τίποτα απολύτως. Αυτά θα πρέπει να συζητούμε εδώ. 24 ώρες μετά από το σκηνοθετημένο δράμα στις ε, Βρυξέλλες γίνεται, συμβαίνει το πραγματικό δράμα, το γνήσιο δράμα και εμείς κάνουμε το κλείνουμε τα μάτια και περιμένουμε να λυθεί το πράγμα από μόνο του. Εδώ χρειάζεται κοινή δράση, εδώ χρειάζεται ενωμένη στάση και να πούμε ξεκάθαρα τα πράγματα με το όνομά τους. Κυρία Ζήμερ, ερώτηση από την κυρία Μαρτέν. Μα με το κύριο, κύριο Μαρτέν, συγγνώμη. Πού βρίσκεστε κύριε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Άκουσα προσεκτικά την κυρία Τσίμε που λέει ότι θα πρέπει να διανεμηθούν οι πρόσφυγες που φτάνουν στην Ελλάδα και αν δεν το κάναμε θα ήταν δραματικό. Γιατί ε, θέλει μόνο στην Ευρώπη αυτή η κατανομή. Γιατί να μην γίνει η κατανομή αυτή στο σύνολο των χωρών, ιδιαίτερα τις γειτονικές χώρες της Ευρώπης. Sehr verehrter η κυρία Γκάβη Αγαπητέ, αξιότιμε κύριε συνάδελφε, είμαστε ευρωβουλευτέ. Είμαστε βουλευτέ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μα έχουν στείλει εδώ οι εκλογέ μα. Βάλουμε στην επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε εδώ. Οι άνθρωποι αυτοί έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είτε το θέλουν αυτοί, είτε το θέλουν άλλοι, ή όχι, είτε το θέλουμε εμεί, είτε όχι, εδώ έρχονται. Δεν αντιμετωπίζονται με κλειστά σύνορα ούτε εξωτερικά κλειστά σύνορα, ούτε εσωτερικά κλειστά σύνορα. Οφείλουμε να έρθουμε στο ύψο των ευθυνών μα. Δεν μπορώ να πάω να πω σε κάποιον άλλον, όχι να του δεχτείτε εσεί. Εμεί έχουμε το κλειδί στο χέρι και εμεί θα πρέπει επιτέλου να ανοίξουμε την κοινή αυτή πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε οι άνθρωποι αυτοί να μπορούν να φτάσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρί να κινδυνεύσει η ζωή του, Να τηρούνται τα προβλεπόμενα από τις συνθήκες για το άσυλο. Ευχαριστώ. Η κυρία Χάρμς, πρόεδρος της ομάδας των Πράσινων. Αγαπητοί συνάδελφοι και εσείς αγαπητοί αγαπητοί σήμερα, βεβαίως η πολιτική πάντα έχει και ένα στοιχείο σκηνοθεσίας. Όμως, στην τελευταία αυτή διάσκεψη κορυφής δεν μου φάνηκε ότι ήταν μονάχα μια φτηνή σκηνοθεσία. Είχα την εντύπωση ότι ο Ντόναλτ Τούσκ σωστά τα περιέγραψε τα πράγματα, ότι ήταν πραγματικά το πέρας μια, μιας πάρα πολύ σοβαρής διαπραγμάτευσης όπου δεν ήταν μοναχά το επίκεντρο αυτή η συμφωνία με τον Κάμερον όπου στο επίκεντρο ήταν η προσπάθεια να πετύχουμε κάτι το οποίο θα μας επιτρέψει να διατηρήσουμε τη συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δική μου εντύπωση, που βεβαίως μόνο ως παρατηρήτρια μπορούσα να την δω την ε, διάσκεψη αυτή, ήταν μια διάσκεψη όπου εν τέλει πολλά από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου έφτασαν στο χείλος του γκρεμού και είδαν πραγματικά ποια είναι η άβυσος που μας περιμένει και τι σημαίνει πραγματικά εάν μια παλαιά μεγάλη χώρα μέλος εγκαταλείψει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελπίζω και το λέω και απέναντι σε όλους αυτούς τους σκυλοκαυγάδες που βλέπουμε να συμβαίνουν στην Μεγάλη Βρετανία. Ελπίζω ότι αυτές οι αντιπαραθέσεις στη Μεγάλη Βρετανία θα βοηθήσουν τους Βρετανούς ψηφοφόρους να διακρίνουν ποιο είναι το όφελος από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ελπίζω ότι όλες και όλοι εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορέσουμε να αντιληφθούμε μέχρι να φτάσει η τελική ψηφοφορία ποιο είναι το όφελος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλο αυτό το οικοδόμημα που έχουμε φτιάξει εδώ και δεκαετίες, όπου έχουν χαθεί και ανθρώπινες ζωές και ειδικά στην Ανατολική Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Όλα αυτά μπορούν να καταστραφούν μέσα σε λίγες εβδομάδες. Μην το λησμονείτε αυτό. Γνωρίζω αρκετά καλά ανθρώπους όπως τυχοδιώκτες, όπως αυτός ο κύριος Φάρατζο απέναντί μου και τι μπορούν να κάνουν. Αυτή η διαδικασία σε βάθος κατανόησης που ανοίγει τώρα στην Βρετανία μπορεί να αποδειχτεί μια διαδικασία που θα μας επιτρέψει σε όλους και όλους να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις. Απέναντι στις κρίσεις των καιρών αυτών, η Ευρώπη μένει όλο και πιο μόνη της, διότι οι Ηνωμένε Πολιτείε και φαίνεται πολύ καθαρά αυτό σε διάφορες συγκρούσεις, δεν θέλουν πια να μας βοηθήσουν να ξεπεράσουμε κρίσεις, αναμένουν από μας και αυτό φάνηκε καθαρά στην Ουκρανική κρίση. Αναμένουν από εμά τι Ευρωπαίε και τους Ευρωπαίους να βρούμε εμείς λύσεις από κοινού. Και αν βλέπω τώρα και τη νέα στατική του Κρεμλίνου απέναντι στη Συρία και αν βλέπω και όλες αυτές τις κρίσεις που οξύνονται ανά τον κόσμο, το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι μαζί με το Ενωμένο Βασίλειο θα μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση καλύτερα να ξεπεράσει την κρίση αυτή με τον ευρωπαϊκό τρόπο. Είναι όμως και το αντίθετο σωστό, ότι και η Μεγάλη Βρετανία θα μπορέσει να αντέξει την κρίση εφόσον βοηθήσει να διατηρηθεί η ενότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι κρίμα που το προσφυγικό έχει αντιμετωπιστεί τόσο φτωχά. Είπατε και εσείς κύριε Γιούνκερ, όταν τα πράγματα δυσκολεύουν τότε ενωνόμαστε. Όμως αυτό δεν το είδα καθόλου εγώ στη διάσκεψη κορυφής στο προσφυγικό. Είδαμε μέσα σε μια αλυσιδωτή αντίδραση και ως συνέπεια της ανικανότητας που έχουμε δείξει απέναντι στο προσφυγικό να υψώνονται ξανά οι φράχτες μέσα στην Ευρώπη και μάλιστα θα τις προστατεύσουν λένε και στρατιωτικά. Το θέμα έχει αναβληθεί για να ξανασυζητηθεί στη διάσκεψη κορυφής με συμμετοχή της Τουρκίας. Εύχομαι σε αυτούς που θέλουν μια πιο δίκαιη πολιτική για το προφέλουν να αντιμετωπίσει οι άνθρωποι δίκαια τους, ή να αντιμετωπίσει η Ένωση τους ανθρώπους αυτούς δίκαια τους πρόσφυγες. Εύχομαι σε αυτούς να δείξουν την μέγιστη διαπραγματευτική ικανότητα. Τα πράγματα θα συνεχίσουν να είναι τα ίδια. Αυτή η κατανομή στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μα κάτι τέτοιο θα έπρεπε να είναι δυνατό. Οι αριθμοί το επιτρέπουν. Καλύτερη διαχείριση των συνόρων. Θα κοστίσει χρήματα αυτό, όμως είναι αναγκαίο και πρέπει να γίνει στην βάση του δικαίου. Το ΝΑΤΟ μπορεί να παρέμβει επικουρικά, δεν μπορεί όμως να ασφαλίσει μόνο του τα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης. Την μεγαλύτερη βοήθεια για τους πρόσφυγες που βλέπουμε στην Ορτανία ή στην Τουρκία διακόπτει ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και για την προσοχή σας και για την υπομονή σας. Κύριε Χάμς, μια στιγμή. Ο κύριος Άρνολτ θέλει να σας, να σας ρωτήσει κάτι. Είστε σύμφωνοι? Εσείς πιστώνετε την Ευρωπαϊκή Ένωση και με πράγματα που δεν έχει κάνει. Κοιτάξτε, για τη συμφωνία. Μιλούμε για μια πιο στενή ενωσία, αλλά αυτό ποτέ δεν βασίστηκε σε τίποτε. Τελικώς παρεξηγείται το πρόβλημα. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι η εξή. Βλέπετε κανένα άλλο συγκεκριμένο παράδειγμα για το τι έχει επιτύχει ο Κάμερον με αυτή τη συμφωνία. No, but sorry, you mentioned απάντηση της κυρία Χάμ στα αγγλικά. Ρωτήσατε ποια είναι η πιο επίγουσα ιδέα. Αυτό το emergency break, αυτό το φρένο ανάγκης. Όμως, εδώ χρειάζεται συμβασμός. Πάντοτε η Ευρώπη βασίζεται στους συμβασμούς. Οτιδήποτε πετύχαμε να προχωρήσει ήταν στη βάση συμβασμού. Ωστόσο, μακροπρόθεσμα. Δεν θα μπορέσω ποτέ να συμφωνήσω εργάτε, για παράδειγμα, που να προέρχονται από ανατολικοευρωπαϊκέ χώρε να θεωρούνται εργάτε δεύτερη κατηγορία. Και ελπίζω ότι τουλάχιστον σε αυτό συμφωνείτε μαζί μου. E για την ομάδα τη Ελευθερία και τη Δημοκρατία έχει το λόγο ο πρόεδρο του, κ. Φάρατσου. Ευχαριστώ. Ήδη είναι αρχικά πάρα πολύ συναρπαστικά είναι εποχή δημοψηφισμάτων. Και στις 6 Απριλίου στην Ολλανδία ξεκινάμε, όπου θα ψηφίσουν για τη συμφωνία με την Ουκρανία και δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι θα το απορρίψουν. Και είπε σήμερα ο κύριος Σόρμα θα γίνει και στην Ουγγαρία ένα δημοψήφισμα για το αν θα πρέπει να τους υποχρεώσουν να δεχτούν υποχρεωτικές ποσοστώσεις για τους μετανάστες μετά από τα μεγάλα σφάλματα της κοινή πολιτικής ασύλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να μην πω και για τις δηλώσεις της κυρίας Μέρκελ. Και ο Τσέχος Πρωθυπουργό λέει ότι υπάρχει αίτηση και στην Τσεχία να υπάρξει ένα δημοψήφισμα για τη συμμετοχή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Α, και στι 23 Ιουνίου θα γίνει το Βρετανικό δημοψήφισμα για το αν θα μείνουμε ή θα φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό οδήγησε σε μια διάσκεψη κορυφή 40 ωρών όπως ο, όπου ο David Cameron έκανε μια ε, παρουσίαση σε στυλ Oliver Twist ζητώντας περισσότερα, περισσότερες παραχωρήσεις και ζητώντας να ακυρώσει τις, ε, ε, τα, τα ωφέλη προς τους μετανάστες για ένα σύντομο διάστημα και επίσης να εξασφαλίσει ότι δεν είμαστε δεσμευμένοι για μια ολοένα στενότερη ένωση. Και θα έχουμε ένα δημοψήφισμα ότι όπου λέει ο Πρωθυπουργό μα ότι θα είναι νομικά δεσμευτική η συμφωνία. Και το είπε και ο κύριο Στάσκ ότι είναι νομικά δεσμευτική αυτή η συμφωνία. Μα είπε ο κύριο Κάμερον όμω, ότι τα έγγραφα αυτά θα τα καταθέσει στα Ηνωμένα Έθνη. Μπορεί να βάλει και τις κάλσες του στα Ηνωμένα Έθνη άμα θέλει, γιατί δεν έχει κανένα απολύτως νόημα να καταθέσει κανείς ένα έγγραφο στα Ηνωμένα Έθνη, μπορεί να τα βάλει σε μια χρηματοθυρίδα αλλά είναι όλα αυτά νομικά δεσμευτικά. Το 2008 είπε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ότι οι υποχρεώσεις οι οποίες προκύπτουν από διεθνές συμφωνίες δεν μπορούν να θίξουν τις συνταγματικές αρχές των συνδικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο σημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο υπεστήριξε τις τωρινές συνθήκες μέχρι να έχουμε μια νέα συνθήκη. Αλλά ποιος λέει ότι θα έχουμε νέα συνθήκη οποιαδήποτε νέα συνθήκη θα οδηγήσει ακόμα περισσότερα δημοψηφίσματα και δεν νομίζω ότι οι μεγάλες ομάδες το κοινοβούλιο θα δεχτούν κάτι τέτοιο. Φυσικά έχουμε και το χειρόφρενο, το φρένο έκτακτης ανάγκης. Αυτό θεωρήθηκε ότι ήταν μια μεγάλη επιτυχία. Αλλά αυτό έγινε μέσα από παράγωγο δίκαιο που μπορεί να ψηφιστεί, που πρέπει να ψηφιστεί από το κοινοβούλιο μας. Δηλαδή θα γίνει δημοψήφισμα. Λέμε μαζί με τον κύριο Κάμερον μένουμε και μετά θα ξαναγυρίσουμε στο κοινοβούλιο. Αυτό το κοινοβούλιο θα υποστηρίξει όμως την στάση των ε, Εγγλέζων που θέλουν να είναι διαφορετικοί από όλους τους άλλους. Από ό,τι άκουσα σήμερα δεν θα γίνει κάτι τέτοιο. Οπότε κύριε Τούς και κύριε Κάμερο, αν με ακούτε, αυτή η συμφωνία δεν είναι νομικά δεσμευτική με κανένα τρόπο. Και πρέπει να σας πω ότι το βρετανικό κοινό θα αποφασίσει τι είναι πιο ασφαλές. Είναι ασφαλές να μείνει με ένα φορέα όπου μας λένε ότι οι αστυνομικέ δυνάμει ότι έρχονται 3 με 5.000, έχουν έρθει 3 με 5.000 τρομοκράτε μέσα από τη διαδικασία μετανάστευση, ή είναι καλύτερο να ξαναπάρουμε τα ενία τη δημοκρατία μα και των συνόρων μα. Σκεφτόμενοι όλα αυτά, εγώ πιστεύω ότι είναι καλύτερο, πολύ καλύτερο για μα να φύγουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Φάρατζ, Υπάρχει ερώτηση από τον Ευρωβουλευτή κύριο Κάσα. Δέχεστε, κύριε Κάσα, εσείς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ξέρουμε ότι ο κύριος Φάραντ θέλει να φύγει το Ηνωμένο Βασίλειο από τότε που ήρθε εδώ. Προσπάθησε με τις τοπικές εκλογές, απέτυχε. Μετά προσπάθησε με τις βουλευτικές εκλογές και εκεί δεν τα κατάφερε και έδωσε μεγαλύτερη πλειοψηφία στον Κάμερον και στο Συντηρητικό Κόμμα. Και τώρα έρχεται ακριβώς ε, το δημοψήφισμα. Στην περίπτωση που πει η πλειοψηφία ναι ε, στο, στην Ενωμένη Ευρώπη, θα εγκαταλείψει επιτέλους την πολιτική ή μήπως θα βρει ακόμα μια ευκαιρία να παραμείνει ανάμεσά μας και να χαρεί και αυτός και εμείς την παρέα του. Κύριε Κάζα, δεν ξέρω ποιος σας ενημερώνει για την εκλογική ιστορία του UKIP, ίσως να μην τα θυμάστε καλά, αλλά το 2014 πήραμε 28% στις ευρωεκλογές σε το σύνολο του Ηνωμένου Βασιλείου αλλάξαμε, ήρθαμε πρώτοι ε, για πρώτη φορά που δεν ήταν το εργατικό ή το συντηρητικό κόμμα πρώτο. Σχετικά τώρα με το δημοψήφισμα, πράγματι νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία ζωής Είμαι βέβαιος ότι αν παραμείνουμε δεν νομίζω ότι θα έχουμε πια καμία ευκαιρία και θα βυθιστούμε βαθύτερα σε αυτή την πολιτική ένωση. Έχουμε όμως την ευκαιρία, η όθηση αυτή τη στιγμή εμείς την κατευθύνουμε, ε, θα ψηφίσουμε υπέρ της αποχώρησης και νομίζω ότι σύντομα όλοι οι ευρωβουλευτές από τη Μεγάλη Βρετανία θα φύγουν και αυτοί. η κυρία Λεπέν από το INF. Κοιτάξτε, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με τις αναλύσεις των εκλογικών αποτελεσμάτων. Ε, ξέρω ότι οι σοσιαλιστές έφτασαν στο 22% στις τελευταίες εκλογές και δεν παρετήθηκε κανείς. Σε τέσσερις μήνες οι Άγγλοι λοιπόν θα αποφασίσουν αν θα μείνουν ή αν θα φύγουν αυτή η λαϊκή κυριαρχία θα είναι μια επιλογή η οποία είναι φυσικά η δείχνει τη δημοκρατική παράδοση του Ηνωμένου Βασιλείου. Ε, τα μέσα ενημέρωσης δεν έχουν όλα την ίδια άποψη, θα γίνει μια πλούσια και δημοκρατική αντιπαράθεση και συζήτηση βλέπουμε την ελευθερία σκέψης, την ελευθερία έκφρασης, τον σεβασμό των διαφορετικών εκφράσεων, η έννοια της δημοκρατίας. Η συζήτηση για το Brexit θα δείξει ποιος είναι ο απολογισμός της συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 70 και μετά. Αν ο απολογισμός δεν είναι ικανοποιητικός θα ακολουθήσουν μια άλλη άποψη, την άποψη της ελευθερίας, της κυριαρχίας η δήλωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του 1793 στο άρθρο 28 εκφράζει μια σαφέστατη αρχή. Μια γενεά δεν μπορεί να επιβάλλει τους νόμους της στις μελλοντικές γενναίες. Μια γενιά των Άγγλων ήθελε η ιστορία η πρόσφατη να εγγραφεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η γενιά αυτή δεν μπορεί να υποχρεώσει τα ευρωπαϊκά όργανα χωρίς ψηφοφορία να επιβάλλονται και για το μέλλον. Αυτή είναι η δημοκρατία και είναι κάτι το απολύτως θεμητό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μας επιβάλλει ολόκληρες σειρές νόμων και αποφάσεων. Αποφάσεις που λαμβάνονται από ανθρώπους που δεν εκλέγονται χωρίς δημοκρατική συζήτηση, χωρίς δημόσιες διαβουλεύσεις, έτσι λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργεί με τυραννικό τρόπο που απέκτησε νόμιμα την εξουσία αλλά ασκεί την εξουσία με καταχρηστικό και επικίνδυνο τρόπο. Και αυτή η συμφωνία και η εφαρμογή της, η ψεύτος συμφωνία και οι εκβιασμοί οι οποίοι πολλαπλασιάζονται από πλευρά του κοινωνικού ε, συστήματος ή ε, φυσικά ε, ε, τα, οι δημοσκοπήσεις του κυρίου Σόρος τους, τις οποίες διαφημίζει ο κύριος Βέμπερ. Μόνο οι λαοί αποφασίζουν. Οι λαοί επενούν, οι λαοί τιμωρούν και αυτό είναι το πνεύμα της δημοκρατίας. Ελπίζω οι κυρώσεις στη συγκεκριμένη περίπτωση, η τιμωρία να είναι βίαιη γιατί οι Βρετανοί θα επιλέξουν την ελευθερία. Η μία εγγεγραμμένη κυρία Ντότς έχει το λόγο. Εμείς στο Ηνωμένο Βασίλειο βλέπουμε την δική μας μέρα ανεξαρτησίας στις 23 Ιουνίου. Το κάνουμε γνωρίζοντας ότι παρά τις καλύτερες προσπάθειες του Πρωθυπουργού μας να επιτύχει την αλλαγή το, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θέλει ούτε μπορεί να φέρει αλλαγή. Η νέα συμφωνία που υποσχέθηκε σε εμά ο David Κάμερον ουσιαστικά έχει χαθεί. Θα συνεχίσει να διαβρώνεται η ανεξαρτησία μας και θα κινδυνεύει η ασφάλειά μας. Θα στέλνουμε περισσότερα εκατομμύρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση από ό,τι παίρνουμε πίσω, δισεκατομμύρια και τα ψεγάδια της συμμετοχής μας θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Ακόμα και εάν δούμε την, ε, τα ψίχουλα τα οποία μας έχουν υποσχεθεί στη συμφωνία δεν υπάρχει καμιά εγγύηση, δεν υπάρχει εγγύηση για αλλαγή των συνθηκών. Δεν μπορεί να το εξασφαλίσει κανείς ούτε αυτό το Κοινοβούλιο ούτε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Έχουμε ενώπιον μας μια παροδία, μια προσπάθεια να πουλήσουν γουρούνι στο σακί στους Βρετανούς. Εγώ θα τους έλεγα μην το αγοράσετε. Θα πρέπει να πιστέψετε στο Ηνωμένο Βασίλειο ο, είπε ένας γνωστός συγγραφέας υπάρχουν πολλά πράγματα μπροστά στο μέλλον από αυτά που αφήνουμε πίσω μας. Έχετε δύο μπλε κάρτες, κυρία Ντότς. Θέλετε να τις δεχτείτε. Από την κυρία Μαγκίνης πρώτα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα μπορούσε η κυρία Ντότς να αναγνωρίσει το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ειρηνευτική διαδικασία στη Βόρεια Ιρλανδία, διότι δημιούργησε χώρο για αυτούς οι οποίοι διαφωνούσαν με την ε, και τους βοήθησε να διαπραγματευτούν. Δεν βλέπετε λοιπόν την αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί υποστήριξε την ειρήνη και ιδιαίτερα στη Βόρεια Ιρλανδία. Δεν μπορούμε προφανώς να παρέμβουμε στο δημοψήφισμα του Ηνωμένου Βασίλειου, εμείς ως γείτονες στο νησί της Ιρλανδίας, πρέπει και εμείς να έχουμε κάποιο λόγο στο θέμα αυτό. Πρέπει να γίνει ακουστή και η δική μας φωνή. Ελπίζω να το δεχτείτε. Να σας ευχαριστήσω κυρία Μαγκίνης. Είναι πράγματι μια πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτησή σας και πάντα αναγνώρισα τον ρόλο τον οποίο αυτό εδώ το Κοινοβούλιο και τα θεσμικά όργανα έπαιξαν στην ειρηνευτική διαδικασία έτσι ώστε να υπάρξουν και πιστώσεις διαθέσιμες για το βόρειο τμήμα της Ιρλανδίας. Πάντως εκτιμάται ότι σε επίπεδο ε, διαφθρωτικών ταμείων ε, ε, όταν παίρνουμε μία λίρα δίνουμε πίσω μία λίρα 58. Οπότε καταλαβαίνετε ότι σήμερα μεν έχουμε καλύτερες σχέσεις διακοινωτικές πολύ καλύτερες από ό,τι στο παρελθόν και θα συνεχίσει ελπίζω η κατάσταση αυτή. Και ελπίζω ότι αυτό θα θεωρεί και ο, ναι, ο κάθε Πρωθυπουργό της χώρας σας. Θέλω οι συζητήσεις να συνεχιστούν, θέλουμε όμως συζητήσεις ειλικρινείς, χωρίς εκφοβισμούς, που ε, δεν είναι υποχρεωτικά κάτι που δεν χαρακτηρίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ενημερώνω ότι εμένω στο προηγούμενο του κυρίου Σούλτς και δέχομαι κάθε φορά μία μπλε κάρτα και γι' αυτό θέλω να δείξετε κατανόηση όσοι έχετε επίσης ζητήσει το λόγο. Περνάμε τώρα στον κύριο Ρόιλ για 1,5 λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εσείς κύριε Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στην τελευταία συζήτηση για την κατάσταση στην Ευρώπη ήμουν μεταξύ εκείνων που επέκριναν το γεγονός ότι στο Συμβούλιο φαίνεται μόνο να συμμετέχουν εγωιστές. Τώρα νομίζω ότι είναι σωστό να πω ότι αυτή εδώ η τελευταία διάσκεψη κορυφής ήταν η απόδειξη του εναντίου. Είμαι πολύ ικανοποιημένος προσωπικά για το γεγονός ότι στην τελευταία διάσκεψη κορυφής επιτέλους το Συμβούλιο κατάφερε να λάβει αποφάσεις έδειξε ότι μπορεί να λύσει πολύ σοβαρά προβλήματα. Ευχαριστώ τον πρόεδρο τους και όλους τους άλλους που συνεργάστηκαν. Δώσατε επιτέλους την απόδειξη ότι η Ευρώπη μπορεί να αναλάβει δράση και στα πιο δύσκολα θέματα. Πολύ σωστά είπε η κυρία Χάρμς ότι όχι μόνο στη Μεγάλη Βρετανία πρέπει να αντιληφθεί ο κόσμος πόσο σημαντικό είναι αυτό το ευρωπαϊκό έργο και εμείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο και στο Συμβουλίο πρέπει να αντιληφθούμε πόσο μεγάλη σημασία έχει αυτό το ευρωπαϊκό εγχείρημα για όλες και όλους εμάς και πού μπορούμε να το προχωρήσουμε με συμβιβασμούς. Εάν γίνει αυτό, τότε έγινε ένα σημαντικό βήμα που ανοίγει νέες ευκαιρίες για την Ευρώπη. Ελπίζω και εύχομαι ιδίω για το θέμα των προσφύγων. Κύριε Φόξ, έχω μεγάλη εκτίμηση στο πρόσωπό σας, αλλά το πρόβλημα το πρόβλημα των προσφύγων στην Ευρώπη δεν οφείλεται στην πρόσκληση μιας καγκελαρίου. Δεν συμφωνώ μαζί σας. Το πρόβλημα είναι τεράστιο και το πρόβλημα λύνεται μόνο με κοινή δράση. Οι αποφάσεις της τελευταίας εβδομάδας μπορούν να αποτελέσουν την αφετηρία για την επίλυση του μεγάλου αυτού προβλήματος. Και δεν θα μπορέσουμε να επιτύχουμε ωστόσο αν δεν συμμετάσχουμε όλοι μαζί στην προσπάθεια αυτή. Ευχαριστώ κύριε Ρόιλ. Κύριε Βίλμοτ, τρία λεπτά. Please. Θα μπορούσαμε να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες της συμφωνίας της προηγουμένης Παρασκευής, αλλά κάτι τέτοιο δεν θα ήταν σωστό. Έχει γίνει η συμφωνία. Συνήφθη η συμφωνία και τώρα το χρονόμετρο προχωρεί. Έδωσαν στον David Κάμερον τη δυνατότητα να ταχθεί επιτέλους σαφώς υπέρ της παραμονής. Ωστόσο, στο δημοψήφισμα δεν θα κριθεί η συμφωνία το ερώτημα που έχουν μπροστά τους οι Βρετανοί πολίτες είναι πολύ πιο σημαντικό από οτιδήποτε μπορεί να συμφωνηθεί σε οποιοδήποτε πρωινό ή πρόγευμα στις ε, Βρυξέλλες. Πρόκειται για το μέλλον της Βρετανίας, αν θα παραμείνει global player ή όχι. Είναι το μέλλον της Ευρώπης. Είναι η στενή διεθνή συνεργασία που χρειαζόμαστε για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του σημερινού κόσμου για υπερβολικά μακροχρονικό διάστημα απέφυγαν οι Βρετανοί πολιτικοί να συζητήσουν τα μεγάλα θέματα της Ευρώπης. Επιτρέψαμε να κυριαρχήσουν στη συζήτηση αυτοί από το απέναντι μέρος του φάσματος. Να διχάσουν τον κόσμο. Να επιβάλλουν τη δική τους ιδεολογική ατζέντα. Αυτοί που λένε μεγάλα παχιά λόγια αλλά δεν δίνουν απαντήσεις όταν τους ρωτά κανείς Ποιε εναλλακτικέ επιλογέ μπορείτε να προτείνετε για να παραμείνει η Μεγάλη Βρετανία δραστήριο μέλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρίε και κύριοι, ήρθε η ώρα να ενισχύσουμε αυτού που είναι υπέρ. Ήρθε η ώρα να ξεβροστιάσουμε αυτού που λένε αυτά τα πράγματα ωστόσο, που δίθεν ισχυρίζονται ότι είναι πατριώτε που οδηγούν όμω σε μια πορεία που θα μειώσουν το παράστημα τη χώρα μα ανά τον κόσμο. Δήθεν τάσσονται υπέρ των εργαζόμενων, ενώ στην πραγματικότητα προωθούν λύσεις που σημαίνουν λιγότερη ασφάλεια για την απασχόληση, λιγότερα κοινωνικά δικαιώματα. Γι' αυτό το εργατικό κόμμα τώρα έχει βγει στους δρόμους και πάει και χτυπάει πόρτες για να εξηγήσει στον κόσμο γιατί πρέπει η Βρετανία να παραμείνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο, άρα να παίξει και πρωτοπόρο ρόλο. Χάρη στην εκστρατεία του Εργατικού Κόμματος και των Συνδικάτων καταφέραμε να εμποδίσουμε τους συντηρητικού να μειώσουν τα δικαιώματα των εργαζόμενων. Εργαζ... Ε, ε, δικαιώματα για, για ισότιμη αμοιβή. Α, όλες αυτές είναι εκστρατείες τις οποίες έχουμε προχωρήσει εμείς. Και θα ταχθούμε υπέρ της παραμονής της Βρετανίας ως ενεργού παίκτη στο παγκόσμιο γίγνεσθε. Να γίνει πιο ισχυρή η Βρετανία σε συνεργασία με τους Ευρωπαίους εταίρους της. Μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα ακόμα για να λειτουργήσει καλύτερα η Ευρώπη εποφελία των εκλογέων μας. Κανείς όμως να μην έχει ε, ψευδεστήσεις. Όταν θα κερδίσουμε το δημοψήφισμα, όταν θα έρθει η σχετική νομοθεσία, δεν θα έχει τελειώσει το έργο μας. Για να μπορέσει να ασκήσει επιρροή στη διαδικασία αυτή η Βρετανία, πρέπει να έχει θέση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Θα αγωνιστούμε με κάθε τρόπο για να κερδίσουμε. Σας ευχαριστώ. Κυρία Βίλμοντ, δέχεστε γαλάζια κάρτα από τον κόμιτα του Ντάρτμπουθ. Uh, Σας ευχαριστώ που δέχεστε την μπλε κάρτα στις βουλευτικές εκλογές εδώ και λίγους μήνες το μανιφέστο του Εργατικού Κόμματος ήταν κατά του δημοψηφίσματος για τον Brexit. Εσείς υποστηρίζετε ε, το δημοψήφισμα ή είστε πάντα κατά. Και αν υποστηρίζετε την τέλεση του δημοψηφίσματος γιατί αλλάζετε γνώμη τότε. Νομίζω ότι δεν έχει σημασία αυτό που λέτε. Έτσι κι αλλιώς είτε μας αρέσει είτε όχι θα έχουμε δημοψήφισμα. Το θέμα είναι εμείς να διασφαλίσουμε το μέλλον του ε, Βρετανικού λαού. Το μέλλον του είναι σε μια ισχυρή Ευρώπη. Αυτό θα βοηθήσει την οικονομία μας, τις επενδύσεις, την απασχόληση και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Η κυρία Ιντβέλτ, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να αναφέρομαι πάντα στη γνωστή τηλεοπτική εκπομπή «Ναι Πρωθυπουργέ μου, Yes Prime Minister». Η ερώτηση ήταν, κοιτάξτε, έχετε τους ίδιους στόχους τα τελευταία 500 χρόνια, να διαιρέσετε την Ευρώπη. Ε, πολεμήσαμε με τους Ολλανδούς εναντίον των Ισπανών, με τους Γερμανούς εναντίον των Γάλλων, με τους Γάλλους εναντίον των Γερμανών και των Ιταλών. Οπότε γιατί να αλλάξουμε τώρα όταν μέχρι σήμερα πήγε καλά το πράγμα. Εγώ σαν Ολλανδή φιλελεύθερη και σαν Ευρωπαία ας αποδείξουμε ότι ο Σερ Χαμφρέι λέει σαχλαμάρες. Αγαπητοί φίλοι, θέλουμε να είστε μέσα στο, στην Ενωμένη Ευρώπη όχι λόγω μιας συμφωνίας λίγο θολής, αλλά γιατί μόνο μέσω μιας ισχυρής Ευρώπης θα ανταποκριθούμε στις προκλήσεις. Πρόσφυγες, τρομοκρατία, οικονομική κρίση, ενεργειακή κρίση και έτσι θα βελτιώσουμε τη ζωή των πολιτών εκμεταλλευόμενοι τις τεράστιες δυνατότητες της ψηφιακής εποχής και της παγκόσμιας οικονομίας. Ναι στο δημοψήφισμα. Ευχαριστώ τώρα η κυρία Άντερσον για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το να σπρώχουμε τους εργάτες πέρα του ορίου ένδυας δεν είναι ο τρόπος με τον οποίο θα μπορέσει να διατηρηθεί το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ψευδής ε, υποσχέση για ανταγωνιστικότητα και σημασιολογικέ τροποποίησεις στην όλο και κοντύτερη στενότερη ένωση δεν θα ικανοποιήσουν τους ευρωσκεπτιστές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βέβαια δεν είναι τέλεια. Είναι μακριά από τους πολίτες, έχει να κάνει με ένα τεράστιο δημοκρατικό έλλειμμα. Είναι μακριά από εκεί που θα έπρεπε να είναι. Και δεν έχει την δύναμη των Εθνικών Κοινοβουλίων, αλλά δίνει ουσιαστική προστασία για τα δικαιώματα των εργαζομένων, των καταναλωτών και για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δίνει ευκαιρίε για τι προοδευτικέ δυνάμει να ενωθούν. <clears throat> Έχει υποστηρίξει την ελλαδική διαδικασία ειρήνευση και προστατεύει τι προσπάθειε για να μειωθεί ο αντίκτυπο των συνόρων με τη χρηματοδότηση για την ε, ειρήνευση, για το ίντερεκ, τις γέφυρες στον Τόνεγκαλ και στον Ταλιχάνα. Πάρα πολλά κονδύλια στον αγροτικό τομέα είχαν τεράστιο αντίκτυπο για την Βόρεια Ιρλανδία και υπάρχουν χιλιάδες πολιτών που <clears throat> δεν έχουν καμιά εμπιστοσύνη στο να αναλάβει αυτό το εγχείρημα η Βρετανική κυβέρνηση μετά από το δημοψήφισμα. Γι' αυτό το Σινφέιν θα αγωνιστεί εναντίον του Brexit. Η θέση της Ιρλανδίας είναι στην Ευρώπη και της Βόρειας και της Νότιας όμως κυρία Ήβανς για ένα λεπτό και 30 δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Για την Ουαλία. Αυτή είναι μια εποχή έντονης πολιτικής συζήτησης. Πριν από το δημοψήφισμα τον Ιούνιο θα έχουμε εκλογές το Μάιο για μια νέα ε, κυβέρνηση και κοινοβούλιο στην Ουαλία. Και μας ενδιαφέρει να μπορέσουμε να φτιάξουμε μια ισχυρή και βιώσιμη οικονομία και να είναι ανθυρές οι κοινότητές μας. Για μένα το μήνυμα αυτό το κόμμα της Ουαλίας πιστεύει ότι η φυσική θέση της Ουαλίας είναι στην Ευρώπη. Εμείς θα αγωνιστούμε για να εξασφαλίσουμε ότι η επιτυχή σχέση μας, η εταιρική μας σχέση με την Ευρώπη θα παραμείνει και στο μέλλον. Είχαμε οικονομικά, πολιτικά, πολιτιστικά και κοινωνικά ε, από την, παροχή, από την παρουσία της Ουαλίας στην Ευρώπη και θέλουμε να συνεχίσουν όλα αυτά. Αλλά αυτό το δημοψήφισμα είναι για τη μεγαλύτερη εικόνα. Είναι για το είδος έθνους που θέλουμε να είναι η Ουαλία και για το είδος ένωσης που θέλουμε να είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση όπου εμείς ως Ουαλοί μπορούμε να συνεργαστούμε και να αναγωνιστούμε τους άλλους για μια καλύτερη κοινωνία. Πιστεύουμε λοιπόν ότι το να παραμείνει η Μεγάλη Βρετανία είναι προ το συμφέρον στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προ το συμφέρον όλων των εργαζομένων μα, όλων των εταιριών μας, του αγροτικού χώρου και κυρίως των νέων της Ουαλίας. Γιατί θα πρέπει να θυμηθούμε ότι αυτή είναι μια ευκαιρία που δεν αφορά μονάχα εμά, αλλά και για τι επόμενε γενιές που θα έρθουν. Ο κύριο Τεχράφ, ένα λεπτό. κύριε Πρόεδρε. Δείχνουν οι δημοσκοπήσεις ότι η πλειοψηφία του βρετανικού πληθυσμού θέλει η χώρα τους να εγκαταλείψει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι δεν έχει την, ε, ε, τη δύναμη να δεχτεί κάτι τέτοιο. Η, προσπάθησε να παραχωρήσει, προσπάθησε να παραχωρήσει πράγματα στους Βρετανούς πριν από το δημοψήφισμα. Αλλά η Βρετανία δεν πρέπει να αποδεχτεί κάτι τέτοιο. Το δημοψήφισμα στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι μια ιστορική καμπή, μια ιστορική ευκαιρία και στις κάτω χώρες. 53% του πληθυσμού θέλει ένα ε, δημοψήσουμε για τη συμμετοχή της χώρας του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελπίζω ότι και αυτό το δημοψήφισμα θα γίνει, ώστε η Ευρώπη να γίνει ένα σύνολο κυρίαρχων κρατών για μεγαλύτερη ευμάρεια. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βόιτ για ένα λεπτό. Σας... Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ακούσαμε σήμερα σχετικά με τα όσα δεν λειτουργούν Ούτε και τα χρήματα για τις υποσχέσεις προς την Τουρκία έχουν συγκεντρωθεί. Ανεξαρτήτως όσα δισεκατομμύρια και να δώσετε στην Τουρκία, η Τουρκία δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα στις συνθήκες. Η Τουρκία έχει συμφέρον να αποσταθεροποιήσει την γείτονά της Ελλάδα, όχι να την βοηθήσει να σταθεροποιηθεί. Ρωτώ λοιπόν, αν αυτό πρόκειται να είναι το ίστατο μέσον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να τα παρατήσει. Ακούσαμε πολλά για το Brexit και για τις καταστροφικές του συνέπειες. Καταστροφικές συνέπειες για την Ευρώπη, για το μέλλον της Ευρώπης. Δεν είναι όμως αυτό. Η έξοδος της Βρετανίας αντίθετα θα φέρει ελπίδα πάλι στην Ευρώπη. Θα διατηρήσουμε ένα πυρήνα της Ευρώπης και θα έχουμε τη δυνατότητα να επιστρέψουμε σε μια Ευρώπη των πατρίδων και των ελεύθερων λαών. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος Πάσκου κυρία Γκροστέτ για ένα λεπτό και 30 δεύτερα. Ευχαριστώ πολύ. Θα πω κάτι το οποίο είχε πει ένας παλιός άλλος πρόεδρος. Έλεγε ότι το σπίτι μας καίγεται, εμείς όμως αποστρέφουμε το βλέμμα, κοιτάμε αλλού, δεν έχουμε τις ίδιες προτεραιότητες. Έγιναν πάρα πολλές συζητήσεις, αλλά δυστυχώς δεν υπήρξαν αποφάσεις για την μεταναστευτική κρίση. Χιλιάδες οι απελπισμένοι που έρχονται στην Ήπειρό μας. Είναι απαράδεκτο, είναι σχρό ε, το εμείς να ασχολούμεθα ε, να αποτρέψουμε το Brexit και να σώσουμε την πολιτική σταδιοδρομία του David Cameron και να ανοίξουμε φυσικά το κουτί της Πανδώρας μιας Ευρώπης à la αυτό θα κοστίσει σε αυτούς που πιστεύουν στην Ευρώπη. Πώς να πείσουμε τους πολίτες ότι μπορούν να προστατευθούν από τα μεταναστευτικά ρεύματα. Μπορούμε να καταπολεμήσουμε τον ΤΑΕΣ, να προστατευτούμε από, τις φτηνές, ε, ε, από τα φτηνά κινέζικα προϊόντα. Νομίζω ότι διάφορες χώρες ε, δημιουργούν προβλήματα στην Ευρώπη η μία μετά την άλλη. Αστάθεια πολιτική, κοινωνική, περιβαλλοντική, στον κόσμο όλο. Απαιτούν από μας να είμαστε ενωμένοι. Θέλουμε εμείς η Ευρωπαϊκή Ένωση να παραμείνει ενωμένη λοιπόν με το Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την Ευρώπη, δεν μπορούμε να κοροϊδεύουμε την Ευρώπη και θα πρέπει επιτέλους τα κράτη-μέλη να μην είναι πυρομανείς αλλά πυροσβέστες. Ευχαριστώ κυρία Γκροστέτ. Κυρία Γκροστέτ. Εάν δέχεστε έχετε μία μπλε κάρτα από τον κύριο Λεμπρετό. Ευχαριστώ που δεχθήκατε την ερώτηση. Λέτε ότι το Brexit θα προκαλέσει περαιτέρω πολιτική και οικονομική αποσταθεροποίηση και μόλις μάθαμε ότι το χρηματιστήριο της Φραγκφούρτης συνήψε μια συμφωνία με το χρηματιστήριο του Λονδίνου. Ε, αυτό δείχνει ότι δεν φοβούνται οι επιχειρηματίες το Brexit και το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να απελευθερωθεί χωρίς καμία βλάβη. Δεν με ακούσατε σωστά, απαντάει η κυρία Γκροστέτ. Εγώ δεν είπα ότι το Brexit θα προκαλέσει πολιτική αστάθεια. Είπα ότι η οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική αστάθεια στον κόσμο απαιτεί από εμά να είμαστε ενωμένοι. Γι' αυτό είναι απαραίτητο 500.000 άνθρωποι, 500 εκατομμύρια μάλλον Ευρωπαίοι να μείνουν ενωμένοι μαζί με το Ηνωμένο Βασίλειο. Όταν βλέπουμε εμείς την κατάρρευση βέβαια του χρηματιστηρίου στο Λονδίνο, νομίζω ότι αυτό που λέτε είναι λάθος. Ο κύριος Γκουερέρο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα δούμε ακριβώς τι θα αποφασιστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο σε τέσσερις μήνες. Ελπίζω να παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρουμε όμως το τι συμβαίνει καθημερινά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά από διαδοχικές κρίσεις, προσφυγικές, κρίσεις ασφαλείας, μετά τη συζήτηση για τον Brexit, ξεχνάμε ότι ζούμε σε μία μόνιμη κρίση εδώ και αρκετά χρόνια μια κρίση απασχόλησης, ανάπτυξης κοινωνικών δικαιωμάτων και χαμηλών μισθών. Ο ΩΣΑ δημοσίευσε τις προοπτικές του τις, επόμενες, τις προηγούμενες εβδομάδες. 1,4 ε, θα αυξηθεί, αναπτυχθεί η ευρωπαϊκή οικονομία, 1 για την Ιταλία, 1,3 για την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε στην κρίση η οποία έχει προκαλέσει εν πολλής και τις άλλες κρίσεις που καταστρέφουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ίσως να φταίνε οι πολιτικές, οι νομισματικές σε, μια, σε ένα πλαίσιο όμως χαμηλού κόστους των πρώτων υλών και σε, με συμφέρουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες. Γι' αυτό ακριβώς επιβάλλει δημοσιονομικές πολιτικές πολύ πιο φιλόδοξες με περισσότερες επενδύσεις και με μεγάλες προοπτικές. Συνεπώς δεν το λέει αυτό μια συνωμοσία κεινσιανών ή κάποιων σοσιαλιστών. Το λέει η κοινή λογική, το λέει η προφανής ανάγνωση αυτών που συνέβησαν τα προηγούμενα χρόνια. Γι' αυτό πρέπει το σχέδιο Juncker να εφαρμοστεί με μεγάλη αποφασιστικότητα και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να αναλάβει περισσότερους κινδύνους σχετικά με, με το προσφυγικό. Το θέμα που συζητάμε είναι ο περιορισμός του, αλλά δεν έχουμε τα μέσα για να αντιμετωπίσουμε αυτό που το προκαλεί. Ο κύριος Γιούνκερ είπε, εγώ άκουσα αυτό που είπε ο κύριος Γιούνκερ σαν κάτι το ηρωνικό. Ελπίζω οι αποφάσεις αυτές κάποτε να εφαρμοστούν. Ευχαριστώ κύριε Γκουερέρο. Μπλε κάρτα από την κυρία Άτκινσον. Σαν σοσιαλιστής, εσείς ε, πιστεύετε αυτά τα οποία λέει ο Κάμερον ε, για Ευρώπη δύο ταχυτήτων. Ε, οι δικοί σας πολίτες από τη μία και όταν έρχονται πολίτες στις χώρες σας από άλλες χώρες όπως η Ρουμανία, Πολωνία κτλ. να αντιμετωπίζονται σαν πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Και όταν έρχονται οι δικοί σας πολίτες μου χώρα να αντιμετωπίζονται εξίσου. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα πρέπει ε, να υπάρχουν τέτοιου είδους καταστάσεις. Εσείς μπορείτε να αποδεχθείτε αυτή την Ευρώπη, εν πάση περιπτώσει, με τις δύο τάξεις πολιτών. Νομίζω ότι η παρέμβαση του υπεύθυνου της κοινοβουλευτικής μου ομάδας όπως επίσης και της κυρίας Βίλμοτ της υπεύθυνη του Εργατικού Κόμματος ήταν σαφής. Εμείς θα υπέρ μιας ισχυρής Ευρωπαϊκής Ένωσης, μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης ολοκληρωμένης και μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία σέβεται όλα τα κοινωνικά δικαιώματα συνολικά και το καθένα ξεχωριστά για όλους τους πολίτες της Ένωσης. Ο κ. Στέλιτσκα για ένα λεπτό. Κυρίες και κύριοι, ερχόμαστε από μια χώρα που ήταν για 40 χρόνια έξω από τη διαδικασία ολοκλήρωσης της Ευρώπης, όχι λόγω της δικής μας θέλησης, αλλά γιατί ήταν το αποτέλεσμα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Υπάρχει τεράστια διαφορά του να είναι κανείς μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το να είναι έξω, παρά τις δυσκολίες, παρά τις ελλείψεις, παρά τις διαφωνίες. Οι Βρετανοί θα πρέπει να το κρίνουν βέβαια. Εμεί όμω θέλουμε το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το χρειαζόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό νομίζω ότι αυτή η συμφωνία που για μένα είναι προβληματική σε πολλά σημεία είναι κάτι που είμαι έτοιμο να το αποδεχτώ και να πληρώσω το τίμημα. Και ένα δεύτερο σημείο που δεν συνδέεται. Αυτό δεν μπορεί να είναι το τέλο όμω. Πρέπει να είναι η αρχή των μεταρρυθμίσεων που χρειάζεται απόλυτα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάποιε από αυτέ είναι τώρα στο επίπεδο των συζητήσεων κάποιε άλλε. Τέλο, προ τον πρόεδρο Τούσκ. Αν δείτε τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και ξέρω ότι κάνετε, μεγάλη προσπάθεια, αυτό δεν είναι επαρκέ. Το Μάρτιο πρέπει να έχουμε κάποια αποτελέσματα ώστε οι πολίτε μα να καταλάβουν και να πιστεύουμε ότι πράγματι κάνουν κάτι για το προσφυγικό. Ευχαριστώ. <clears throat> Ο κύριος Φλάναγκαν για ένα και μισό λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Είναι εκατομμύρια πολιτών Ιρλανδικής καταγωγής θα ψηφίσουν στο δημοψήφισμα του Brexit. Ελπίζω να ακούσουν αυτό που έχω να πω και να κρίνουν ε, από τις απαντήσεις που θα μου δοθούν. Ο κύριος Γιούνκερ, ο οποίος δεν <clears throat> άδειασε να είναι στην ε, Ολομέλεια, του ζητήθηκε να μειώσει το βάρος, να ακυρώσει το βάρος των 31 δισεκατομμυρίων που, που επευλήθηκε στην Ιρλανδία. Διαδοχικές κυβερνήσεις της Ιρλανδίας αναγκαστήκανε να δεχτούν χρέος το οποίο θα μπορούσε να είχε αποφευθεί. Δεν απάντησε όμως ο κύριος Γιούνκερ. Από τότε υπάρχει, έκτοτε υπάρχει τώρα μία ε, προσφυγή ενός μέρους του Κοινοβουλίου στο ανώτατο δικαστήριο της Ιρλανδίας σε σχέση με την νομιμότητα αυτών των οφειλών που δέχτηκε η Ιρλανδία. Ουσιαστικά θεώρησε το δικαστήριο ότι αυτά δεν ήταν δάνεια αλλά ήταν κεφάλαιο των τραπεζών που πήγε και ότι δόθηκαν χρήματα σε μια τράπεζα που ήταν αφαιρέγγια για να την διασώσουν. Και αυτό έγινε δεκτό από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα γιατί φοβόταν την επιμόλυση και την διάδοση της κρίσης. Κύριε ε, Γιούνκερ με τον τρόπο αυτό υποχρέωσε την Ιρλανδία να δώσει 20 δισεκατομμύρια περισσότερο από ό,τι είχαν μαζεύσει σε φόρους το 2010. Θα το δεχόταν η Γερμανία, θα το δεχόταν η Γαλλία. Γιατί δεν απαντάτε σε αυτό το ερώτημα. Αυτό το οποίο καταλαβαίνω εγώ είναι ότι δεν δίνεται πεντάρα και θα, με τον τρόπο αυτό λέω στους Ιρλανδούς να ψηφίσουν υπέρ της αποχώρησης της Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κυρία Σκότια, μισή λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συγγνώμη, δεν είδα την μπλε κάρτα του κυρίου Τάνοκ. Δέχεστε την μπλε κάρτα του κυρίου Τάνοκ. Κύριε Φλάναγκαν. Δέχεστε την μπλε κάρτα από τον κύριο Τάνοκ. Κύριε Τάνοκ. Με μικρόφωνο παρακαλώ. Με μικρόφωνο οι Βρετανοί που ζουν στη χώρα μου εμένα μου φαίνεται πολύ παράλογο αυτό που λέτε. Δεν ξέρω πώς θα βοηθήσετε εσάς και την Ιρλανδική Δημοκρατία να αντιμετωπίσει τα ελλείμματα του τραπεζικού συστήματος. Θέλετε και η δική σας χώρα να φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να γίνει κομμάτι του, ε, του Ηνωμένου Βασιλείου και της ζώνης της Τερλίνας. Αυτό μου λέτε και λέτε ότι αν φύγουμε θα υπάρχει τελωνιακό σύνορο μεταξύ της Βόρειας Ιλλανδίας και της ε, Δημοκρατίας της Ιλλανδίας που θα θέσει περισσότερο βάρος στη Δημοκρατία της Ιλλανδίας. Και πώς αυτό λοιπόν θα βοηθήσει τις θέσεις εργασίες και την ευμάρεια στην ε, Νότια Ιλανδία όταν υπάρχουν σύνορα τα οποία θα επιβάλλουν δασμούς. Και η χώρα σας θα είναι ακόμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Όλα αυτά είναι ηρωνικά γιατί είπα ότι οι Ιρλανδοί δεν έχουν γίνει ακουστοί. Εσείς ακούσατε παρόλα αυτά αυτά που είπε ένα Ιρλανδός βουλευτής. Αυτό που είπα ότι αν δεν έχουμε πραγματικές απαντήσεις σε όλα αυτά γιατί μας κλέψανε τρεις φορές μισό δισεκατομμύρια ευρώ εφέτος που χάθηκαν. Αυτό το οποίο λέω είναι ότι αν ο Ιρλανδικός λαός που δεν τον ακούει κανένας θα πρέπει να καταλάβουν αυτοί που είναι στη Μεγάλη Βρετανία, κάποιοι από αυτούς που έζησαν την κρίση, κάποιοι από αυτούς που ήταν οι κοσάριδες. 205.000 άνθρωποι φύγαν από την Ιρλανδία τα τελευταία πέντε χρόνια. Αν δεν πάρουμε μια απάντηση, το μόνο συμπέρασμα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μας ακούει καθόλου. εκτός αν φέρνει δεξιές πολιτικές, ακροδεξιές πολιτικές όπως τη μετανάστευση. Ευχαριστώ, λέει η κυρία Κότ. οι πράσινοι θέλουμε η Βρετανία να μείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί θέλουμε να εργαστούμε για κοινέ λύσει συλλογικέ προκλήσει που έχουμε ενώπιόν μα. Η ρήπανση των ωκεανών, η κλιματική αλλαγή, οι πρόσφυγε και οι τρομοκράτε δεν έχουν καμία σχέση με τα σύνορα που πρέπει να αντιμετωπιστούν με συνεργατικέ και πλήρε λύσει. Μέχρι τώρα η συζήτηση για το αν το μέλλον μα είναι στην Ευρώπη ή όχι κυριαρχείται από μεσήλικέ ανθρώπου που φοράνε κοστούμια. Αλλά αυτό είναι ίσως το πρώτο κομμάτι, το ντοκιμαντέρ πριν από την ταινία. Τώρα όλοι έχουμε το ίδιο δικαίωμα να αποφασίσουμε. Εγώ συμμερίζομαι τις απόψεις αυτών που νομίζουν ότι η ευρωπαϊκή πολιτική έχει ξεπεράσει αυτά που θέλαν οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου και άλλων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω όμως παρόλα αυτά ότι θα πρέπει να καταλάβουμε την επιτυχία του ευρωπαϊκού χειρήματο όταν άνθρωποι από διάφορε προελεύσει και κουλτούρε εργάστηκαν όλοι κοινοί για το ευρωπαϊκό κοινό καλό. Δεν είναι τέλεια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να μείνουμε μέσα για να την βελτιώσουμε. Είναι μια ευκαιρία να συζητήσουμε για το πώς μια διαφορετική Ευρώπη είναι εφικτή. Ας δούμε πώς μπορούμε να περιορίσουμε την επιρροή των μεγάλων πολυεθνικών και πώς μπορεί να γίνει η Κομισιόν πιο δημοκρατική και να λογοδοτεί στους πολίτες της Ευρώπης. Είναι μια ευκαιρία για να έχουμε μια Ευρώπη των λαών και για τους λαούς. Κύριος Βιλίνσκι για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, πρώτα εκφράζω την χαρά μου διότι στις 23 Ιουνίου στη Μεγάλη Βρετανία θα γίνει μια πραγματικά δημοκρατική πράξη και οι άνθρωποι θα μπορέσουν εκεί να αποφασίσουν πραγματικά τι επιθυμούν. Και στην Ολλανδία τάσεται μια μεγάλη πλειοψηφία υπέρ της διεξαγωγή δημοψηφίσματος. Και στη δική μου χώρα, την Αυστρία, υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι λοιπόν, γιατί να μην είναι δυνατόν στην Ήπειρο εκείνη, όπου γεννήθηκε η δημοκρατία, είτε, είτε γεννήθηκε στην Ισλανδία, είτε γεννήθηκε στην ε, ε, Ελλάδα, αυτά να τα δουν ιστορικοί. Αλλά στην Ήπειρό μας, γιατί να μην επιστρέψει η δημοκρατία. Τι καλύτερο πράγμα υπάρχει, τι πιο δημοκρατικό υπάρχει σε σε οποιοδήποτε δημοκρατικό σύστημα, η πλειοψηφία του κόσμου είναι αυτή. Αυτός είναι ο κυρίαρχος. Ο κυρίαρχος είναι ο λαός. Και έτσι θα κάνει ένα βήμα μπροστά η Ευρώπη, εάν μπορέσει να βάλει τους ανθρώπους μέσα στο δημοκρατικό γίγνεσθε, στο δημοκρατικό παιχνίδι και όχι ανάποδα. Ευχαριστώ. Κορυμπή και ένα λεπτό. Όταν ο Ντόναλτ Τάσκ είπε ότι θέλει να αντιμετωπίσει το, το προσφυγικό πρόβλημα, ξέχασε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι τμήμα του Σέγγεν. Φοβάμαι ότι χρειαζόμαστε μια κοινή οικονομία, αλλά δεν χρειαζόμαστε μια ομάδα ύποπτη ε, επισήμων και πολιτικών που λαμβάνουν αποφάσεις για όλους χωρίς να έχουν το δικαίωμα. Ελπίζω λοιπόν το Ηνωμένο Βασίλειο να φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να επανέλθει στην ΕΖΕΣ. Και ελπίζω επίσης και η Τσεχία και η Σλοβακία και η Πολωνία. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να καταστραφεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Κόρβιν Μίκε, θέλετε μία μπλε κάρτα από τον κύριο Μπονάνο. Eh, Άκουσα αυτά τα οποία είπε ο συνάδελφος. Θα ήθελα να του πω, αν είχε ένα μαγικό ραβδί, αν ήταν στη θέση του Τούσκ ή του Γιούνκερ, τι θα έκανε. Το πρώτο πράγμα που θα έκανε, τι θα ήτανε. repeat your question, the second part of your question. What, what I would do if what? Τι θα έκαναν συνέβαινε τι. Αφού άκουσα την παρέμβαση του κυρίου Κόρβιν Μίκε, αυτό που είπατε δηλαδή, αν είχατε ένα μαγικό ραβδί, αν ήσασταν εν πάση περιπτώσει ένας μάγος, και αν αύριο ε, ήσασταν στη θέση του Ιούνκερ ή στη θέση του Τούσκ. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνατε για την Ευρώπη. Θα έλεγα ότι τελείωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα κοίτα το τέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευτυχώς ζούμε στον πραγματικό κόσμο, λέει ο πρόεδρος. Ο κύριος Γκονθάλες Πόνς για 1,5 λεπτό με χωρίς μικρόφωνο ο μιλητής. Κύριε Πρόεδρε, η συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι αυτό το οποίο θέλαμε, αλλά ήταν η μόνη δυνατή λύση. Κάναμε ό,τι μπορέσαμε για να μην τα χάσουμε όλα. Δεν πρέπει όμως να θεωρούμε ότι είναι μια καλή είδηση. Είναι μια υπαναχώρηση. Η γενιά που έζησε τους δύο παγκοσμίους πολέμους και τις συνέπειές της εξαφανίζεται. Είναι όλο και λιγότεροι Ευρωπαίοι που θυμούνται τις αιτίε και τις συνέπειες του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτό είναι επικίνδυνο. Θέλουμε να έχουμε μια Ευρώπη για να, έχουμε περαιτέρω, να μην έχουμε περαιτέρω εθνικές αντιπαραθέσεις και αυτή τη στιγμή χειροκροτούμε τους ηγέτες που χρησιμοποιούν τις αντιπαραθέσεις αυτές για να έχουν μεγαλύτερη δημοτικότητα. Η Ευρώπη δεν δημιουργήθηκε με ένα πόλεμο έγινε για να μην γίνει πόλεμος στο μέλλον. Δεν πρέπει να την διαλύσουμε μέσα στις αντιπαραθέσεις και το λαϊκισμό. Μιλήσαμε πολύ για τους εξωτερικούς κινδύνους, η πραγματική κίνδυνη για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εσωτερική κίνδυνη. Όπως ήταν και το 1939 οι παλιοί εθνικισμοί και οι παλιοί εθνικισμοί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το μόνο εμβόλιο που έχουμε για να αντιμετωπίσουμε τον πόλεμο. Ας μην την αποδυναμώσουμε. Χρειαζόμαστε το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά η Ιρλανδία, η Αγγλία, η Σκοτία και η Ουαλία μαζί ή από κοινού χρειάζονται πολύ περισσότερο την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει πολύ κρύο. Και κάτι ακόμα θέλω να σας πω. Θα γίνει το δημοψήφισμα. Οι Βρετανοί θα πούν αν λένε ναι ή όχι. Αλλά σας λέω κάτι και πρέπει να το υπενθυμίσουμε. Η Ευρώπη ανεξάρτητα από τους Βρετανούς θα συνεχίσει και θα συνεχίσουμε να μιλάμε για το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά δεν θα υπάρχουν Άγγλοι στην αίθουσα. για δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, η συμφωνία στην οποία καταλήξαμε ομόφωνα, όλες οι 28 εννοώ χώρες, είναι μια δίκαιη και ισορροπημένη συμφωνία. Νομίζω ότι όλα τα θεσμικά όργανα πρέπει να είναι υπερήφανα γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση μπόρεσε εγκαίρως να καταλήξει κάπου. Η συμφωνία αναγνωρίζει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα εξακολουθεί να χρησιμοποιεί και να ωφελείται από την ενιαία αγορά χωρίς να δεσμεύεται από την ολοένα πιο ολοκληρωμένη Ευρώπη ενώ η αρχή αυτή παραμένει πλήρως ενισχύ για τις άλλες χώρες. Η Συμφωνία ε, δίδει εγγυήσεις ε, εναντίον των διακρίσεων και είναι συμβατή με τις συνθήκες και με την ανάγκη διατήρησης ενός πεδίου ε, δίκαιου στο εσωτερικό της ενιαίας αγοράς. Αναγνωρίζει η Συμφωνία την ανάγκη τέρο ολοκλήρωση της Ευρωζώνης Γι' αυτούς τους λόγους, εάν οι Βρετανοί πολίτες αποφασίσουν να παραμείνουν στην Ένωση, τότε θα εξετάσουμε τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με, με υψηλά επίπεδα σεβασμού και δεν θα αποτρέψουμε και ούτε θα καθυστερήσουμε την εφαρμογή των προτάσεων αυτών. Σε επίπεδο νομικό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μόνον τυπικά μπορεί να πάρει μέρος στη διαδικασία αυτή επί τη βάση της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αλλά σε πολιτικό επίπεδο η συζήτηση δείχνει ότι νομίζω ότι η συμφωνία αυτή την χάνει τη στήριξη της πλειοψηφίας του σώματος. Θα είμαστε δίκαιοι, θα τηρήσουμε το λόγο μας και θα πρέπει και οι Βρετανοί πολίτες να διατηρήσουν την ευμάρειά τους στο μέλλον. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Μπέρντερ. Ε, ευχαριστώ τους ε, Ευρωπαίους ηγέτες για την ανοχή τους απέναντι στις απαιτήσεις ε, των συντηρητικών και του κυρίου Κάμερον. Έχει ξεκινήσει η μάχη για το δημοψήφισμα, δεν έχει κερδιθεί ακόμα. Δυστυχώς διάφοροι κομικοί χαρακτήρες όπως ο κύριος Φαράζο και ε, κάποια μέσα ενημέρωσης ε, υπερβολικά έχουν δημιουργήσει μια στρεβλή εικόνα. Πρέπει να παραμείνει το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ευρώπη. Είναι η πρόσβαση στην ευρύτερη ενιαία αγορά ε, Νομίζω ότι είναι και πολύ περισσότερο είναι το θέμα της αντιμετώπισης των κλιματολογικών αλλαγών, ε, της τρομοκρατίας, ε, το μεταναστευτικό και δεν θα πρέπει εμείς να κρυβόμαστε από την πραγματικότητα. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει ε, βοηθώντας ο ένας τον άλλο να βοηθήσουμε τις μελλοντικές γενιές. Ευχαριστώ. Η κυρία Σαρτζεντίνη, ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που οργανώνετε ε, συνέχεια διασκέψη κορυφής με την Τουρκία, χωρίς την Τουρκία, με την Ελλάδα, χωρίς την Τουρκία, με την Αυστρία, χωρίς την Αυστρία, με τις Βαλκανικές χώρες, χωρίς τις χώρες των Βαλκανίων, χωρίς την Ελλάδα, με την Αυστρία και τα Βαλκάνια δεν έχει σημασία αλλά δεν μπορούμε με όλα αυτά να ελέγξουμε την κρίση των προσφύγων αν αρκούμαστε να κατανοήσουμε το γεγονός ότι το 2015 έχουν έρθει ένα εκατομμύριο στην Ευρώπη και θα έρθει άλλο ένα τουλάχιστον αυτή τη χρονιά. Αντί να μιλάμε για τα εσωτερικά και τα εξωτερικά σύνορα, αποστρέφουμε τα ομάτά μας. Οι Υπουργοί Δικαιοσύνη και Εσωτερικών αυτό θα κάνουν όταν μιλήσουν για την ανάγκη να χρησιμοποιήσουν ένα διαφορετικό άρθρο της συνθήκη του Σέγγεν για να κλείσουν τα σύνορα και πάλι λιγάκι. Θα πρέπει να δώσουμε μια θέση στους πρόσφυγες και όχι απλώς να θεωρούμε υπεύθυνε στην Τουρκία και την Ελλάδα. Ευχαριστώ. Έχετε μια πλεκάρτα από την κυρία Βάτσεμπεργκ. Εντάξει. Πρόσεξα προσεκτικά άκουσα αυτά που είπατε κυρία Σαρτζεντίνη. Για σας το πρόβλημα του προσφυγικό οφείλεται στις συνόδους κορυφής στις οποίες αναφερθήκατε ή στο γεγονός ότι δεν υπάρχει βούληση όλα τα κράτη-μέλη να συμφωνήσουν με τις αποφάσεις της μετεγκατάστασης αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση να ασκήσει μια πιο πιεστική πολιτική στην Τουρκία να συμφωνήσει στις υπογραφές που έχει βάλει για επανεισδοχή των οικονομικών μεταναστών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η κρίση δεν αφορά μόναχα τους μετανάστες. Υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι είναι πρόσφυγες και πρέπει να τύχουν καθεστώτους ασύλου. Εγώ νομίζω ότι είναι θέμα πολιτικής θέλησης, πολιτικής αμφασιστικότητας. Η απάντηση του να είμαστε πιο αυστηρή για την Τουρκία δεν είναι μια απάντηση. Δεν έχουμε ε, πληρώσει ακόμα τα 3 δισεκατομμύρια. Δεν θέλουμε να ανοίξουμε άλλα κεφάλαια, δεν θέλουμε να γίνουμε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν θέλουμε να έχουν τη δυνατότητα να ταξιδεύουν χωρί βίζα. Παρ' όλα αυτά θέλουμε να μείνουν τα 2,5 εκατομμύρια εκεί. Αυτό δεν είναι ακριβώ καλή διαπραγμάτευση. Ο κ. για ένα λεπτό διεύθυνση που προηγήθηκε δεν με έπεισε στο ότι είναι κακό το να μπορούν να αποφασίζουν οι Βρετανοί πολίτες αν μείνουν ή αν φύγουν. Και νομίζω ότι δείχνει η κατάσταση ότι το Συμβούλιο δεν αποφάσισε τίποτα το ουσιαστικό ε, για τη μετανάστευση. Έδωσε δώρο τρία δι στην Τουρκία για να εντατικοποιήσει τους ελέγχους. Να θέσω λοιπόν κάποιες ερωτήσεις προς την Επιτροπή κυρίως και τον Πρόεδρο κύριο Τούσκ. Υπάρχει ένας Ευρωπαίος πολίτης ο οποίος ε, συνελήφθη, βασανίστηκε, ε, ο Ρετζένη, και η Ευρώπη η οποία ασχολείται με τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν τολμά να, να, να μιλήσει. Είναι ντροπή αυτό που έγινε. Θέλουμε να ξέρουμε από την Αίγυπτο τι ακριβώς έγινε, πότε θα μας πούν την αλήθεια. Έχει ζητηθεί αυτό από την Ιταλική κυβέρνηση. Αλλά πού είναι η Ευρώπη, πού είναι η φωνή της Μογκερίνη. Είναι απούσα η Ευρώπη και είναι ντροπή αυτό που γίνεται. Ο κύριος Φουντούλη σε ένα λεπτό. Το πρόσφατο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο απέδειξε πως το οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει κανένα μέλλον με την παρούσα μορφή. Κάποια στιγμή σύντομα οι εξελίξεις θα τρέξουν πολύ γρηγορότερα από όσο μπορεί να αντιδράσει ο δυσλειτουργικός αυτός οργανισμός. Η Βρετανία απαιτεί ειδικό καθεστώς εάν και εφόσον παραμείνει στην Ένωση, διότι με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζει τα συμφέροντα των πολιτών της και την εθνική της κυριαρχία. Όμω και άλλε χώρε θα έπρεπε να δικαιούνται να επιτύχουν το ίδιο. Βεβαίω τα κράτη μέλη αλλά και η ίδια η ένωση εύκολα υπέκυψαν μπροστά στι απαιτήσει του ηνωμένου βασιλείου αλλά λίγο καιρό πριν στραγγάλισαν την ελλάδα εξαναγκάζοντας το λαό τη σε φτωχοποίηση. αυτό όμω δεν είναι ούτε ισότιμη μεταχείριση ούτε ευρωπαϊκή αλληλεγγύη ούτε κανένα άλλο από τα ψέματα πάνω στα οποία έχει οικοδομηθεί αυτή η ένωση σχετικά με τα υπόλοιπα συμπεράσματα του συμβουλίου όσο και αν σας ικανοποιεί η έλευση του νάτο στο αιγαίο να γνωρίζετε πως ο ελληνικός λαός θεωρεί την κίνηση αυτή ως προδοσία τόσο εκ μέρους της κυβέρνησης όσο και εκ μέρους των δίθεν συμμάχων μας οι οποίοι χαϊδεύουν την τουρκία ένα κράτος χορηγό των τρομοκρατών που δεν έχει καμία θέση στην ευρώπη. κάντε όσα σχέδια θέλετε για συνδιαχείριση του αιγαίου για τη μετατροπή τη Ελλάδα σε αποθήκη λαθρομεταναστών οι έλληνες πολύ σύντομα θα δώσουν την πρέπουσα απάντηση στα σχέδιά σας. Mr. 1 minute and 30 seconds. λεπτό. Κύριε Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και εσείς κύριε Επίτροπε, ευχαριστώ τους κύριους Τούσκ και Γιούνκερ για την εξαιρετική συνεργασία που πρόσφεραν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη διάρκεια της διασκέψης κορυφής. Νομίζω ότι δεν πουλήσαμε την ψυχή της Ευρώπης και τα συμφέροντά της και η Μεγάλη Βρετανία έλαβε τα δέοντα για να μπορέσει να προχωρήσει στο δημοψήφισμα. Δεσμευτήκαμε ότι θα διατηρήσουμε την ανεξαρτησία του νομοθετικού έργου αλλά ότι θα οδηγήσουμε σε πέρας με κοινή προσπάθεια το έργο αυτό. Και νομίζω ότι αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι και, και αυτό έδειξε μάλλον και η ατμόσφαιρα στις διαπραγματεύσεις. Πιστεύω ότι η συμφωνία είναι στεγανή και νομικά. Και χρειαζόμαστε βεβαίω τη σχετική νομοθεσία να έρθει μετά στο τραπέζι του Κοινοβουλίου. Και θα μπορέσουμε να εκπληρώσουμε αυτό που είπε ο Ντέβιτ Κάμερον και στο τέλο των διαπραγματεύσεων. Και η Μεγάλη Βρετανία σε αυτόν τον αλλαγμένο κόσμο δεν έχει καμιά ευκαιρία να αντιμετωπίσει ούτε τον αγώνα κατά τη τρομοκρατία ούτε τίποτε άλλο μόνη της έξω από την Ευρώπη. Όταν βλέπουμε τώρα τις μέρες αυτές ότι Αμερικανοί και Ρώσοι προχωρούν σε συμφωνία χωρίς εμάς, αυτό επιτέλους πρέπει να μας ξυπνήσει. Είτε όλοι μαζί είτε αλλιώς έχουμε χάσει το παιχνίδι. Ελπίζω ότι η συμφωνία που επιτάφθηκε στη διάσκεψη κορυφής θα ενισχύσει το ρεύμα των Βρετανών ψηφοφόρων υπέρ της παραμονής της χώρας τους. Θα δεχθείτε μια γαλάζια κάρτα, μόνο μία, κύριε Μπρόκ, από τον κύριο Άντερσον. Κύριε Άντερσον, ευχαριστώ. Κύριε Μπρόκ, πιστεύω ότι μια συμφωνία που δεν αναγνωρίζει το ηθικό δικαίωμα των χωρών εκτός της Ευρωζώνης να από το αποτυχημένο πείραμα του ευρώ, πείραμα του ευρώ της λυπεί κάτι. Δεν συμφωνείτε ότι σε αυτό θα πρέπει κάποια στιγμή να συμπληρωθεί η συμφωνία. Μα κοιτάξτε, λέει καθαρά η συνθήκη της Λισαβόνας ότι 26 χώρες μέλη έχουν αναλάβει τις σχετικές υποχρεώσεις. 19 τις έχουν εκπληρώσει, οι υπόλοιπε αναμένουν. Υπάρχει μια διαφοροποίηση. Μόνο δύο χώρες διαθέτουν opt-out για την υπόθεση της Ευρωζώνης. Έχουμε διατηρήσει τη σταθερότητα της εξέλιξης του ευρώ. Έχουμε συμφωνήσει ότι θα εμβαθυνθεί η Ευρωζώνη. Βεβαίως όλοι έχουν τα ίδια δικαιώματα και παίζουν σε πεδίο ισότιμου ανταγωνισμού οι χώρες, οι υπόλοιπες χώρες θα προσχωρήσουν στην Ευρωζώνη. Έχουμε πει ότι δεν υπάρχει, δεν θα υπάρχει ευρωπαϊκή ζώνη με πολλαπλά νομίσματα. Το ευρώ είναι το νόμισμα της Ευρώπης. Κύριε σε ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, αναφερθήκατε για τις επενδύσεις και για το Σέγγεν. Νομίζω ότι αυτά είναι μια πολύ καλή ιδέα. Γιατί η τωρινή κατάσταση κατακαιρματισμού της περιοχής του Σέγγεν απαιτεί κατεπίγουσα δράση και πρέπει να προστατεύσουμε τα ευρωπαϊκά σύνορα. Τι είναι όμως τα πραγματικά ευρωπαϊκά σύνορα. Δεν πρέπει να είναι ένας φράκτης με σειρματόπλεγμα ώστε να έχουμε ένα φρούριο Ευρώπη πίσω από το φράκτη αυτό. Στον 21ο αιώνα εμείς θα πρέπει να έχουμε την Ευρώπη όχι ως φρούριο αλλά ως ένα σύνολο που μπορεί να οργανώσει καλύτερα τη σχέση του με τους εταίρους τους, ώστε τα πραγματικά ευρωπαϊκά σύνορα θα πρέπει να είναι η προχωρημένη υποδομή με επιμελητία, με συλλογή πληροφοριών, ώστε να υπάρχει η ασφάλεια για τους Ευρωπαίους πολίτες να διαχειριστεί τις ροές και να δώσει βοήθεια στους ε, πρόσφυγες. <clears throat> θα πρέπει να είναι λοιπόν μια μεγάλη επένδυση για το μέλλον και αυτή η επένδυση θα πρέπει να αποφασιστεί πολύ σύντομα. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό κύριε Άτκινσον. Έχουμε κάποιους ε, πολίτες μου, εκλογής μου από την Νοτιοανατολική Αγγλία και καλώς ήρθατε. Ελπίζω σας αρέσει η συζήτηση. Ο Ντέβιτ Κάμερον πήρε το 1% μονάχα αυτού που ήθελε και όχι καμία αλλαγή στις ε, συνθήκες. Ήμουνα παρούσα στην ε, συνέλευση των Προέδρων μαζί με τον κύριο Μπρόκ. Αλλά εκπροσωπούμε πάρα πολλούς Βρετανούς που λένε αυτό το οποίο πρέπει να λεχθεί, ότι δεν πρέπει να πιστεύουμε ότι θα υπάρξει περιορισμό στην ελεύθερη κυκλοφορία, δεν θα αναλάβουμε πάλι τον έλεγχο των συνόρων, το λεγόμενο emergency break, το φέρνο ασφαλείας, θα διαμφισβητηθεί ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Επομένω, κύριε Μπροκ, η συμφωνία των Πρωθυπουργών δεν αξίζει το χαρτί το οποίο, στο οποίο είναι γραμμένο. Και το είπε ο Μάικλ Γκόβ, ο Υπουργό Δικαιοσύνη τη Μεγάλη Βρετανία. Ο μόνο τρόπο για να υπάρξει πραγματική ε, αλλαγή είναι να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να πούμε έξω. Κυρία Σόιντροβα, μισή λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε αγαπητοί φίλοι, και εγώ θα ήθελα να καλωσορίσω την πρόταση αυτή. Είναι μια συμφωνία η οποία εκφράζει την επιθυμία 27 χωρών κάτω από συνθήκες αποδεκτές και από το Ηνωμένο Βασίλειο και από τις υπόλοιπες χώρες. Είναι λογικές οι προτάσεις αυτές. Θα πρέπει βέβαια να μην ξεχνάμε ότι η συμφωνία αυτή στην ουσία απαιτεί συζητήσεις για νομικές αλλαγές που και αυτές θα συζητηθούν εδώ. Νομίζω ότι η κόκκινη γραμμή είναι οι κοινέ μας αξίες που δεν θα επιτρέψουν στην αλλαγή των συνθήκων. Λοιπόν, πρέπει να καταπολεμήσουμε την πολεμική ε, και ε, την ε, λαϊκιστική ρητορική. Χαίρομαι που άκουσα τον κύριο Φόξ να ομιλεί υπέρ της παραμονής του Ηνωμένου Βασιλείου και από την άλλη βέβαια ο κύριος Φαράζ παρερμήνευσε τον Τσέχο Πρωθυπουργό. Τι είπε ο Τσέχος Πρωθυπουργός ότι αυτό θα μπορούσε αν φύγει το, ή το Ηνωμένο Βασίλειο να δημιουργήσει αρνητικές επιπτώσεις ε, για αντίστοιχα φαινόμενα άλλων χωρών. Δεν θέλουμε εμείς να φύγουμε από το Ηνωμένο Βασίλειο. Αν όμως ε, ε, υπάρξει ένα όχι στο δημοψήφισμα τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Είμαι επίσης υπέρ της ενέργειας που επέδειξε ο κύριος Τούσκος στις διαπραγματεύσεις. Κυρία Γκραπίνη, ερώτηση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ θα συμφωνήσω ότι το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να παραμείνει εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και νομίζω ότι και εσείς το ίδιο επιθυμείτε. Θα ήθελα λοιπόν να θέσω την εξής ερώτηση. Μετά από τις παραχωρήσεις οι οποίες έγιναν από το Συμβούλιο προς το Ηνωμένο Βασίλειο και εφόσον υπάρξει ναι στο δημοψήφισμα, εσείς πιστεύετε ότι η ελευθερία διακίνησης και οι κανόνες της ε, ενιαίας αγοράς θα γίνουν σεβαστοί. Είμαι πεπισμένη ότι η συμφωνία θα είναι μια καλή για όλους συμφωνία, θα σεβαστεί τις αξίες και τους κανόνες της ε, ενιαίας αγοράς. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά σε επίπεδο νομοθετικό, αλλά οι βασικές αρχές δεν θα πρέπει να παραβιαστούν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι ορθό που έχουμε τώρα βάση για να διεξαχθεί το δημοψήφισμα στην Μεγάλη Βρετανία. Είναι σωστό και είμαι βέβαιος ότι οι Βρετανοί ψηφοφόροι θα λάβουν τη σωστή απόφαση. Δυστυχώς αναλύθηκαν άλλες σημαντικές αποφάσεις σχετικά με το προσφυγικό που για την ώρα μας απασχολεί ως γνωστόν σοβαρότατα. Είναι κρίμα που αναβλήθηκε η απόφαση για την 5η Μαρτίου. Είναι η τελευταία ευκαιρία που θα έχουμε και χρειαζόμαστε επιτέλους ενίσχυση των υποδομών στις χώρες προελεύσεως. Χρειαζόμαστε περισσότερη ασφάλεια στα σύνορα που δεν μπορούμε να αποκαταστήσουμε φράζοντας τα εσωτερικά σύνορα. Χρειαζόμαστε ενίσχυση της Ελλάδας και για την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων και είναι αναγκαίο επιτέλους να στήσουμε στα πόδια της μια πραγματική ευρωπαϊκή λύση. Το έδειξε αυτό και έρευνα που έκανε το Ίδρυμα Μπέρτελσμαν. Φάνηκε καθαρά από τι απαντήσει των ερωτωμένων ότι ήρθε η ώρα της ευρωπαϊκής λύσης και όχι ο καθένας μόνος του. Κύριε Κάρας, Κύριοι Πρόεδροι, κύριε και κύριοι, και τα δύο θέματα, και το προσφυγικό και το ζήτημα του Βρετανικού δημοψηφίσματος έχουν ωστόσο ένα κοινό στοιχείο. Δηλαδή ότι υπάρχουν πολλοί πολιτικοί άνδρες που συνδέουν, που τους λείπει αξιοπιστία, που παίζουν με τους φόβους και τις ελπίδες των ανθρώπων αντί να ψάξουν να βρουν λύσεις. Και τα δύο θέματα αυτά έχουν το κοινό στοιχείο ότι υπάρχουν άνθρωποι και από τα δικά μας πολιτικά στρατόπεδα που προσπαθούν να λύσουν τα ενδοκομματικά τους προβλήματα αλλά και να τονώσουν το δικό τους προφίλ σε βάρος της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, σε βάρος του ευρωπαϊκού εγχειρήματος. Απευθύνω έκκληση προς όλες και όλους σας. Σταματήστε αυτό το παιχνίδι. Τα πράγματα είναι υπερβολικά σοβαρά και στο ζήτημα του προσφυγικού αλλά και στο ζήτημα του Βρετανικού δημοψηφίσματος αυτό που παίζει το σημαντικότερο ρόλο είναι η ενότητα της Ευρώπης. Όχι επανεθνικοποίηση, όχι προβολή των εθνικών εγωισμών. Αυτά πρέπει να λεχθούν γρήγορα και καθαρά. Είναι απαράδεκτο. Η, η παραβίαση του δικαίου αφενός να δικαιολογεί παραβίαση του δικαίου από τον άλλο. Είναι απαράδεκτο φράχτες από εδώ ε, να δικαιολογούν φράχτες από εκεί. Το διεθνές δίκαιο, το ευρωπαϊκό δίκαιο, οι αξίες μας, οι αποφάσεις που διαθέτουμε είναι επαρκείς για να επιτρέψουν μια κίνηση προς μια ξεκάθαρη λύση και προς τη μια αποκατάσταση της αξιοπιστίας. Κύριε Κάλλας, μια γαλάζια κάρτα από τον κύριο Μπαλτσίτης ε, Κύριε Αρτουή. Με συγχωρείτε, λέει ο πρόεδρος, με συγχωρείτε αγαπητέ κύριε. Με συγχωρείτε κύριε, με συγχωρείτε, λείπουμε πολύ. Τον λόγο έχει λάβει ο κ. Μπαλτσίτης, διότι ζήτησε πρώτος, λείπουμε πολύ. Ο κ. Μπαλτσίτης. αγαπητέ Κάρας. Είπατε πολλά. Ορισμένοι από εμά θεωρούμε όντως ότι η Μεγάλη Βρετανία πρέπει να παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να θριαμβεύσει η λογική. Δεν θεωρείτε όμως ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να θεσπίσει μέτρα για την περίπτωση όπου η Μεγάλη Βρετανία δεν θα αποτελεί πλέον τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν πρέπει να αρχίσουμε να μιλούμε για το City του Λονδίνου και για άλλα πράγματα. Να συζητήσουμε για αυτά, να είμαστε έτοιμοι για οποιοδήποτε ενδεχόμενο. Οι διαπραγματεύσει των τελευταίων ημερών, ευχαριστώ και όλες και όλους που τα συζητήσατε τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ τον Έλμαρ Μπροκ, Κουτιέρε Βερχόφστατ, όλα τα πρόσωπα αυτά, ευρωβουλευτές, οι οποίοι συνέβαλαν ώστε να υπάρξει συμφωνία, γιατί με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ώστε μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δράσει η Ευρώπη ως μια ενότητα και όχι να θυσιαστεί αυτή η Ευρωπαϊκή Ενότητα στον βωμό των εθνικών εγωισμών. Ο Μάνφρετ Βέμπερ αναφέρθηκε στους πολίτες που ελπίζουμε ότι θα ενισχύσουν την ενότητα. Στο δημοψήφισμα δεν θα ψηφιστεί η συμφωνία, θα ψηφιστεί ναι ή όχι η παραμονή της Μεγάλης Βρετανίας. Ωστόσο αυτό που πρέπει να υπάρξει είναι η συμπαράταξη. Σας ευχαριστώ και Κάρας. Λόγω της παρανοήσεως προηγουμένως νομίζω ότι είναι δίκαιο ε, να ε, επιτρέψουμε κατ' στον κύριο Ατουή να θέσει την ερώτησή του αν δέχεστε κι εσείς. Μάλιστα, βεβαίως. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Καράς. Να σας ε, ομολογήσω ότι μου επετέθησαν πολύ όταν τόλμησα να πω ότι η συμφωνία των κρατών μελών με τον κύριο Κάμερον ήταν επιτυχία. Γιατί αυτό δίνει την εντύπωση μιας πολιτικής αδυναμίας. Λες και η Ευρώπη έχει έλλειψη ηγετικής ε, θέσης, ηγετικής ε, δύναμης και ικανότητας να δράσει. Αυτά τα οποία ζητούνται από τον Βρετανικό λαό δεν θίγουν το ευρωπαϊκό όραμα. Δεν έχουμε λοιπόν μία τέτοια αντιμετώπιση. Εγώ θεωρώ ότι αυτή η συμφωνία ανοίγει την πόρτα σε όλες τις ε, διεκδικήσεις. Δεν θα μπορούμε να κάνουμε τίποτα για τέσσερις μήνες για αυτό το δημοψήφισμα το οποίο μπορεί να μην γίνει. Πάλι υπάρχουν κοινά στοιχεία στα θέματα. Υπάρχουν αποφάσεις. Υπάρχει όμως και μια έλλειψη σοβαρότητας σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των αποφάσεων. Και αυτό βαρύνει αυτούς που έλαβαν τις αποφάσεις. Αυτοί πρέπει οι ίδιοι να πάρουν σοβαρά, στα σοβαρά τον εαυτό τους. Και αν αυτό δεν συμβεί, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Το ίδιο λοιπόν ισχύει για το προσφυγικό, όπως και για τη συμφωνία με το Ενωμένο Βασίλειο. Ξαναλέω, στο δημοψήφισμα δεν θα ψηφιστεί η συμφωνία, παρά το ναι ή όχι παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ αναμένω από τους πολιτικούς αυτούς να δείξουν σοβαρότητα και να προχωρήσουν στην, στις συζητήσεις και στις διαπραγματεύσεις με σοβαρό τρόπο. Να στηρίξουν τα όσα έχουν πει και τα όσα έχουν συμφωνήσει και να τα φέρουν μέχρι τέλους. Νίτερ Μιούλερ, ένα λεπτό mindenkinek az az érdeke hogy az egyesült királyság az európai unió része maradjon. mégis a meg... Παρ' όλα αυτά η συμφωνία αυτή, εφόσον την ε, διαβάσει κανείς προσεκτικά, δεν μπορεί να είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένος, ιδιαίτερα λόγω της μείωσης. Θέλει αυτό, έχει ένα διακριτικό χαρακτήρα. Αφήνει μια πικρή γεύση στο στόμα μας, γιατί ο κύριος Φάρας και η άκρα δεξιά ήταν αυτοί που ξεκίνησαν αυτή την εκστρατεία εναντίον των εργαζομένων από την Ανατολή. Ξέρουμε ότι οι Ούγγροι και οι Πολωνοί δεν πηγαίνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο λόγω των κοινωνικών επιδομάτων. Το κάνουν επειδή δεν έχουν δουλειά στη χώρα τους. Το να μην έχουν κοινωνικά επιδόματα σημαίνει ότι αυτοί δεν θα μπορούν να βλέπουν τις οικογένειές τους. Αυτό μας αφήνει μια πικρία, γιατί για μια ακόμα φορά τους αναγκάζουμε να πληρώνουν αυτοί για μια σύγκρουση στην οποία αυτοί δεν έχουν καμία σχέση. Είναι οι πιο ευάλωτοι. Με τον τρόπο αυτό θίγουμε περισσότερο τους φτωχούς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όταν υπάρχει μια σύγκρουση, η πρώτη λύση είναι ας, κάτω, ας κόψουμε τις κοινωνικές παραχές. Πάντα αυτή είναι η λύση που προτιμάμε και τώρα έχουμε κράτη-μέλη τα οποία θέλουν να κάνουν κάτι τέτοιο. Εγώ θέλω να αγωνιστώ για μια Ευρώπη η οποία δεν ενδιαφέρεται μόνο να περικόπτει κοινωνικές δαπάνες. Κυρία Σούιτσα, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Έχουμε φτιάξει μια Ευρωπαϊκή Ένωση για να μην έχουμε συγκρούσεις και πολέμους και να έχουμε ειρήνη. Όχι όμως για να υποκύπτουμε στο λαϊκισμό. Αυτοί που δημιούργησαν αυτή την Ένωση ήταν αρκετά θαραλέοι για να έχουν τη ζώνη του Σέγγεν, την Ευρωζώνη, για να ενώσουν την Ευρώπη. Πρέπει να το διατηρήσουμε αυτό. Ο πρόεδρος Βέμπερ είπε και σωστά ότι στον πόλεμο της Λιβύης, στην Ουκρανία, στη Συρία εμείς δίνουμε δεν δώσαμε αρκετή σημασία γιατί δώσαμε σε προτεραιότητα το Brexit, το Brexit. Μα είναι μια πραγματική προτεραιότητα στις κρίσεις που αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα με την ανεργία που είναι τόσο ψηλή στις χώρες μας. Ο κύριο Γιούνκερ είπε πρόσφατα ότι είτε θα είμαστε θαραλέοι ή όλα θα καταρρεύσουν. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε θαραλέοι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να καταρρεύσει και πιστεύω ότι ο λαός του Ηνωμένου Βασιλείου θα είναι αρκετά λογικός και θα κάνει τις σωστές αποφάσεις τον Ιούνιο. Πιστεύω θα πούνε ναι και θα παραμείνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι το μόνο σωστό και για την Ένωση και για το Ηνωμένο Βασίλειο. Είπατε κύριε Τάσκ και σας ευχαριστώ ότι είναι μια από τις πιο δύσκολες και επικίνδυνες στιγμές στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι σωστό. Αλλά συγχρόνως βρισκόμαστε μέσα στα πλαίσια μιας τεράστιας ανθρωπιστικής και προσφυγικής κρίσης, μεγαλύτερης από το Δεύτερο Παγκοσμίο Πόλεμο. Γι' αυτό περιμένω από την 7η, 7 Μαρτίου με αδημονία γιατί ελπίζω ότι θα υπάρξουν κάποια αποτελέσματα από τη διάσκεψη κορυφής με την Τουρκία και τότε δεν θα χρειαζόμαστε άλλες συζητήσεις. Προτού σας ρωτήσω αν δέχεστε ή όχι την μπλε κάρτα από τον κύριο Γιάκοψης. πρέπει να σας πω ότι θα ζητήσουμε από την κυρία Γκυγιόμ να λάβει το λόγο και μετά θα ακούσουμε τον πρώτο γιατί πρέπει να φύγουμε, να φύγει και μετά συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Αυτό είναι το σενάριο. Δέχεστε την κάρτα του κύριου Γιάκοφτσιτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κυρία Σουίτσα που δέχεστε την μπλε μου. Εγώ άκουσα με μεγάλη προσοχή, σας γνωρίζω, γνωρίζω ότι θέλετε το Ηνωμένο να παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εγώ το ίδιο νιώθω. Αλλά δεν θα αποφασίσουμε εμεί, ούτε θα αποφασίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο Βρετανικό λαό θα αποφασίσει. Αν ο Βρετανικό λαό αποφασίσει ότι θέλει να φύγει, δέχεστε ότι αυτή είναι η ουσιαστική απάντηση του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν πρέπει να προκύψουν περαιτέρω διαπραγματεύσεις. Τότε, αν θέλει να ξαναμπεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να αρχίσει διαπραγματεύσει από την αρχή. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στο ερώτημά σα. Ναι, συμφωνώ μαζί σα ότι η συμφωνία η οποία έχει γίνει είναι οριστική. Αλλά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει κάνει παραχωρήσει, έχει ψηφίσει ομόφωνα για το θέμα αυτό και δεν νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε στους Βρετανούς την ευκαιρία να αναδιαπραγματευτούν την παραμονή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η απάντηση είναι ναι, λοιπόν, σε αυτό που με ρωτήσετε. Η κυρία Γκυγιόμ, για το θέμα αυτό του Brexit και των προσφύγων, το ίδιο ερώτημα βρίσκεται από πίσω. Μπορεί να μείνει ενωμένη στην πολυμορφία και στις, στα δύσκολα η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχουμε μια στρατηγική για τα προσφυγικά, αλλά τι αποφασίστηκε απολύτω τίποτα. Αυτό το οποίο έγινε ουσιαστικά είναι να εγκριθεί κάτι το οποίο έπρεπε ήδη να ισχύει, αλλά στην πράξη επιτοπίως δεν είχε εφαρμοστεί. Αυτή τη στιγμή η η Ιταλία και η Ελλάδα είναι υποχρεωμένες να φέρουν όλο το βάρος. Και επίσης υπάρχουν μονομερείς αποφάσεις που λαμβάνονται δεξιά και αριστερά. Ο ένας θέλει μια ποσόστοση για τους πρόσφυγες, ο άλλος θέλει να επιλέγει τους πρόσφυγες στα σύνορά του. Έχουμε μια Ευρώπη η οποία όλο και περισσότερο είναι στην απομόνωση. Όλο και περισσότερο όπως στην περίπτωση της Ελλάδος γιατί η αλυσίδα που περνά από τις χώρες των Βαλκανίων έχει τήξει περισσότερο την Ελλάδα, το σπάσιμο της αλυσίδας. Δεν μπορεί λοιπόν το Συμβούλιο να αντιμετωπίσει την πραγματική ανθρωπιστική κρίση. Θέλουμε λοιπόν να πολλαπλασιάσουμε τι ευρωπαϊκέ διασκέψει κορυφή χωρί να παίρνουμε αποφάσει. Δεν πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για λόγου πολιτική προπαγάνδα την προσφυγική κρίση. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ο πρόεδρο του έχει το λόγο. Και μετά ο επίτροπο κ. Τομπρόφσκι στο τέλο. Ευχαριστώ πολύ για την κατανόηση που επιδεικνύεται. Υπάρχουν δύο θέματα τα οποία συζητάμε σήμερα. Το θέμα του Ηνωμένου Βασιλείου και το θέμα της μετανάστευσης συνδέονται μεταξύ τους. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο τρόπος που θα αντιμετωπίσουμε το θέμα της μετανάστευσης θα έχει πολύ μεγάλη σημασία και για την εκστρατεία για το δημοψήφισμα. Όσοι θέλουν να διατηρηθεί η ενότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ενότητα της Δύσης και όλοι αυτοί οι οποίοι φοβούνται ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε τεράστιες δυσκολίες πρέπει να επιδείξουν την μέγιστη δυνατή αποφασιστικότητα και ένα κοινό πρόγραμμα μια ουσιαστική εφαρμογή των αποφάσεών μας με πλήρη σεβασμό των ρυθμίσεων του Σέγγεν και με κοινή δράση με την Τουρκία. Αυτή η διαφαινόμενη κοινότητα δράσης ε, στα προσφυγικό, αν παραβιαστεί από οιονδήποτε, τότε θα συνεισφέρει στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως είπα, η ρύθμιση για το Ηνωμένο Βασίλειο θα τεθεί σε λειτουργία εφόσον ο Βρετανικός λαός αποφασίσει να παραμείνει. Αν ψηφίσει να αποχωρήσει, τότε η συμφωνία πάβει πλέον να υπάρχει. Και κανένας δεν θα πρέπει να έχει αδίποτε ψευδέστηση σε αυτή την περίπτωση. Δεν ήταν ένας από τους διάφορους γύρους των διαπραγματεύσεων, ήταν ο πρώτος και ο τελευταίος. Δεν θα υπάρξουν πλέον τέτοιες ευκαιρίες. Σας ευχαριστώ, συγγνώμη, αλλά για λόγους τεχνικούς πρέπει να αποχωρήσω πλέον. Ευχαριστώ κύριε Τούσκ. Τώρα θα δώσω στον κύριο Κεφαλογιάννη το λόγο για 1,5 λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, δύσκολα κανείς μπορεί να διαφωνήσει με τις οποθετήσεις του κυρίου Γιούγκερ και του κυρίου Τούσκ για δίκαιη συμφωνία με τα ευρωπαϊκά κράτη και το ηνωμένο βασίλειο. αν βγει όχι από το δημοψήφισμα δεν υπάρχει άλλη διαπραγμάτευση. το ηνωμένο βασίλειο η μεγάλη βρετανία όπως την ονομάζαμε για πολύ καιρό η ομιλία του Ίσον Τσόρτζη το 1947 στη Ζηρίχη που πρώτος μίλησε για τις Ηνωμένε Πολιτείες της Ευρώπης η θέληση των λαών της Σκωτίας, της Ουαλίας, της Βόρειας Ιρλανδίας γεννούν ένα ερώτημα. Αυτό το δημοψήφισμα διακινδυνεύει για το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Μεγάλη Βρετανία να γίνει η μικρή Αγγλία, περιθωριοποιημένη στην Ευρώπη και στον κόσμο. Μεταναστευτικό. Επενδύομαι στην ενίσχυση της Σέγγεν. Επενδύομαι στην προστασία των ευρωπαϊκών συνόρων και όχι στο κλείσιμο των ευρωπαϊκών συνόρων. Η Τουρκία είναι μέρος του προβλήματος αλλά και μέρος της λύσης εξισώνει το μεταναστευτικό με την ενταξιακή της πορεία αφήνει ανεξέλεγκτους τους παράνομους διακινητές δέχεται χωρίς βίζα όλους τους πολίτες των χωρών της βόρειας αφρικής δεν εφαρμόζει το πρωτόκολλο επανεισδοχής δεν δέχεται πίσω κανένα από τους παράνομους πρόσφυγες. όλοι μαζί με ευθύνη και σοβαρότητα θα πρέπει να βρούμε λύσεις. είμαι βέβαιος ότι η ευρώπη και θέλει και μπορεί και είναι σε θέση να το επιτύχει. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Το Κένγκε για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εμείς παρακολουθήσαμε μια ακόμη συνάντηση κορυφής που δεν καταλήγει πουθενά και που παραπέμπει σε μελλοντικές αποφάσεις. Αυτό δείχνει το βάθος της κρίσης της Ένωσης. Για να αντιμετωπίσουμε τη μεταναστευτική κρίση, στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είναι ο περιορισμός των προσφυγικών ροών και η αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης. Νομίζω ότι αυτά δεν τα έχει καταφέρει ακόμα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Όταν θέλει κανείς να διαχειριστεί ένα τέτοιο φαινόμενο πρέπει να διασφαλίσει ασφαλείς τρόπους μετανάστευσης και πρέπει να ενσωματώσει τους μετανάστες στον κοινωνικό και οικονομικό ιστό της χώρας, της κάθε χώρας. Ε, το σχέδιο έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το μεταναστευτικό φαινόμενο δίδει κάποιες πρώτες απαντήσεις. Νομίζω ότι έτσι θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε με μεγαλύτερη αλληλεγγύη και με ανάληψη ευθύνης. Νομίζω ότι από πλευράς Ευρώπης πρέπει να δούμε μακριά, γιατί αλλιώς θα αποτύχουμε πολιτικά και θα απαγορεύσουμε και την ελεύθερη διακίνηση των πολιτών. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χέκμαρκ, μισή λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, είναι εντυπωσιακό ότι στις ε, σημερινές συζητήσεις λίγες από αυτές στράφηκαν γύρω από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Εδώ δεν είναι θέμα μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς θέλουμε να εξελιχθεί. Μιλούμε για την Ευρώπη, για τη σταθερότητα, την ειρήνη, την ε, ανάπτυξη βλέπουμε από τη μια μεριά Πούτιν, Ρωσία, Ουκρανία. Προκλήσεις απέναντι σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες μέλη. Πολλοί από αυτούς που μίλησαν από εκεί θα ήθελαν να υποχωρήσουμε απέναντι στον Πούτιν. Έχουμε ωστόσο την ανάγκη για οικονομική ανάκαμψη, ευημερία. Και από τούτην δω την πλευρά που δείχνω δεν θέλουν ανοιχτές αγορές. Όμως αν εξετάσουμε τα προβλήματα πραγματικά σχετικά με τη σταθερότητα. Όπως είπα, ο Πούτιν, η κατάρρευση χωρών στη Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική, η κρίση του προσφυγικού, οι πολιτικές για την προστασία του κλίματος, δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς, οποιοδήποτε να ισχυριστεί ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά χωρίς ενότητα. Και αυτοί που επιζητούν τον κατακαιρματισμό στηρίζουν μόνο τις προσδοκίες του Πούτιν, των Λεπέν και ούτω καθεξής. Πρέπει να τους νικήσουμε αυτούς. Πρέπει να κατανοήσει και το ίδιο το ΕΒ πόσο σημαντική είναι η θέση του στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Κύριε Χέκμαρκ, υπάρχει μια γαλάζια κάρτα από τον κύριο Γιούρεκ. Συμφωνείτε να δεχτείτε να απαντήσετε. Αυτό που θα με εξέβλητε ήταν να μην θέλει κανείς να με ρωτήσει κάτι. Κύριε Γιούρεκ, 30 δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για αυτά που είπατε για τον ρόλο της Ρωσίας στην Ευρώπη, ιδίως στο τμήμα της Ευρώπης, το οποίο βρίσκεται η δική μου χώρα. Αλλά βλέπετε ότι δεν είναι οι πολίτες οι οποίοι θέλουν να συζητήσουν την κρίση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι οι κυβερνήσεις και ομάδες πίεσης που αποδέχονται τέτοιες πρωτοβουλίες όπως το Nord Stream 2 που είναι επικίνδυνες για τη χώρα μου και τη δική σας χώρα. Α μην θεωρείτε λοιπόν ότι οι χώρε και η κοινή γνώμη φταίνουν. Ας κινητοποιήσουμε τους λαούς και τις κυβερνήσεις. 30 δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ. Είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι ο λαό της Ευρώπης δίνει προτεραιότητα στην σταθερότητα και την ασφάλεια του τμήματος του κόσμου μας. Θέλουν ασφάλεια και βλέπουν τις απειλές. Θέλουν να έχουμε μια ενεργειακή πολιτική που να είναι υπεύθυνη και μια πολιτική προσφυγική που να είναι υπεύθυνη. Πρέπει να εξασφαλίσουμε εμεί ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά και να δείξουμε το δρόμο. Και δεν πιστεύω ότι κάποιο θεωρεί ότι μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα αυτά καλύτερα με το να κινηθούμε μόνοι μας. Παρακαλώ κλείστε. Ευχαριστώ. Η επόμενη ομιλήτρια είναι η Έλενα Βαλεντιάνο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Έχουμε δώσει πολύ χρόνο στο να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε, να αποτρέψουμε την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι κάνουμε πολύ καλά με το να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε τον Brexit. Με, με εκπλήσει όμως ο λίγος χρόνος και η λίγη προσπάθεια που έχουμε αφιερώσει στο να ε, αποτρέψουμε την ευρωέξοδο, δηλαδή την έξοδο των κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις αξίες και τις αρχές που θα πρέπει να είναι η βάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε την κρίση των προσφύγων. Η κρίση των προσφύγων είναι η πραγματική κρίση αυτή τη στιγμή της Ευρώπης αυτή τη στιγμή. Αυτού που η Ευρώπη έχει διεκδικήσει να κάνει και που ήθελε να είναι. Όλα αυτά είναι κάτι που θέτει ένα αμφιβόλο όλα αυτά που έχουμε υποστηρίξει στο παρελθόν. Ενώ λοιπόν έχουμε εργαστεί για να αποφύγουμε το Brexit, έχουμε ξεχάσει ότι πρέπει να αποφύγουμε την ευρωέξοδο, την εξαφάνιση των αρχών της δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης που είχε μέχρι τώρα εκπροσωπήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά τώρα πια όχι. Ευχαριστώ. Ο τελευταίος ομιλητής είναι ο κύριος ε, Ρανζέλ πριν από τη διαδικασία κάτι για 1,5 Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για μένα τα αποτελέσματα αυτού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σε ό,τι αφορά το θέμα του Ηνωμένου Βασιλείου και τις συμφωνίες που επετέθη, είναι ικανοποιητικά τα αποτελέσματα. Εγώ θεωρώ ότι <clears throat> μπορέσαμε να διατηρήσουμε τις θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε κάποιες από τις ε, αιτήσει του Ηνωμένου Βασιλείου και γι' αυτό είχαμε μια προσέγγιση θέσεων η οποία ήταν ισορροπημένη, ήταν ισορροπημένη και είναι αποδεκτή. Αυτό το οποίο για μένα είναι το αποφασιστικό σε αυτό το θέμα είναι το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία βέβαια δεν πρέπει να παρέμβει καθόλου στην κυρίαρχη θέληση του Βρετανικού λαού, που θα πρέπει να αποφασίσει με κάθε ελευθερία αν θέλει να παραμείνει ή αν θέλει να φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να κάνει απόλυτα σαφή τη θέση μας. Ότι αν η επιλογή είναι η έξοδος της Μεγάλης Βρετανίας, αυτό θα είναι ανεπίστρεπτο. Θα πρέπει να το γνωρίζουν και οι Ευρωπαίοι πολίτες και κυρίως οι Βρετανοί πολίτες ότι υπάρχουν πλέον εκτήματα και μειονεκτήματα και καλά θέματα και, καλά, και κακά με το να είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν και δικαιώματα και υποχρεώσεις. Θα πρέπει λοιπόν να είναι απόλυτα σαφές ότι δεν θα υπάρξει δεύτερη διαπραγμάτευση και θα πρέπει να επομιστούν όλες τις επιπτώσεις της εξόδου της χώρας τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με όλα αυτά η απόφαση του Βρετανικού λαού και οποιοδήποτε άλλο λόγο θα πρέπει να είναι κυρίαρχη και ελεύθερη. Η διαδικασία Catch the Eye τώρα. 14 ομιλητές έχουν ζητήσει το λόγο. Μέχρι 10 μπορώ να του δεχτώ αλλά θα πρέπει να παραμείνετε μέσα στα πλαίσια του ενός λεπτού. Θα με διευκολύνετε για να δώσω το λόγο σε όλους. Κύριε Μακίνες, ένα λεπτό. Um, Ευχαριστώ πολύ. Η, το Συμβούλιο συζήτησε τα θέματα της μετανάστευσης. Αλλά όλη η συζήτηση μας σχεδόν είναι για το Βρετανικό δημοψήφισμα. Θα ήθελα να ξεκινήσω να μιλήσω για αυτό το θέμα της μετανάστευσης, γιατί συνδέεται με αυτά που γίνονται στο Ηνωμένο Βασίλειο και το ενδεχόμενο αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει κάνει αρκετά. Αν δείτε τι έχει κάνει η Τουρκία, ο Λίβανος και η Ορδανία, που έχουν κάνει μεγάλες προσπάθειες και έχουν πάρει υποσχέσει χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν έχουν πάρει ακόμα τα χρήματα αυτά. λοιπόν είναι ένα θέμα που χρειάζεται μεγαλύτερη προσπάθεια και μεγαλύτερη εστίαση, γιατί Όλα αυτά οδηγούν σε αρνητική θέση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το θέμα του Ηνωμένου Βασιλείου μίλησα ήδη προηγουμένω. Δεν πρέπει να παρεύουμε καθόλου, αλλά έχουμε τη δυνατότητα να εκφράσουμε τη γνώμη μας και εγώ ω γείτονα του Ηνωμένου Βασιλείου, ω Ιρλανδί και με την Βόρεια Ιρλανδία στα σύνορά μας, εμείς θέλουμε να έχουμε κάποιο συμφέρον να διατηρηθεί το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Καπούτο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Απαντώντας στην μεταναστευτική κρίση δέχτηκε το Συμβούλιο την προσφορά του ΝΑΤΟ στον έλεγχο των παράνομων κινήσεων στο Αιγαίο. Η πλήρης εφαρμογή του προγράμματος δράσης με την Τουρκία είναι θα έλεγα μια τεράστια προσπάθεια για να περιοριστούν οι μετανάστες. Πρέπει να περιορίσουμε τον αριθμό αυτό και με άλλες προσπάθειες και άλλα μέτρα έτσι ώστε να εφαρμοστεί σωστά το πρόγραμμα δράσης. Απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για να πετύχει η προσπάθεια και η συνάντηση κορυφής της 7ης Μαρτίου είναι καθοριστική. Για το Brexit νομίζω ότι ε, θα πρέπει να φανούμε πάρα πολύ προσεκτικοί έτσι ώστε να μην είναι κάτι το μοιραίο για την ευρωπαϊκή οικονομία και για την οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου. Πρέπει να παραμείνει το Ηνωμένο Βασίλειο περισσότερη Ευρώπη για να σωθεί η Ευρώπη. Ο κύριος Μαριάς για Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε οι τούρκοι δουλέμποροι συνεχίζουν να στέλνουν χιλιάδες πρόσφυγες στην ελλάδα τα σκόπια συνεπικουρούμενα από την αυστρία κλείνουν τα σύνορα με αποτέλεσμα η ελλάδα να κινδυνεύει να μετατραπεί σε ένα απέραντο προσφυγικό νταχάου ενώ η γαλλία η γερμανία η δανία η αυστρία η σουηδία και σήμερα το βέλγιο έχουν αναστείλει τη σέγγεν. η υποκρισία γύρω από τη μετεγκατάσταση συνεχίζεται αφού από τις 66.400 πρόσφυγες που δεσμεύτηκε η ευρωπαϊκή ένωση να πάρει από την ελλάδα δεν έχουν μετεγκατασταθεί ούτε 400 η ελλάδα όσο παραμένει στη σέγγεν αποτελεί μαγνήτη για τους χιλιάδες πρόσφυγες μια και τους χορηγεί ταξιδιωτικά έγγραφα τύπου σέγγεν που τους επιτρέπουν να ταξιδεύουν στη γερμανία. γι' αυτό διακινδυνεύουν οι πρόσφυγες να πνιγούν στο αιγαίο αντί να πάνε από τη ε, βουλγαρία προς τη γερμανία. μόνη λύση η ελλάδα να αποχωρήσει από τη σέγγεν να κλείσει τα σύνορά της και να αναθέσει τη φύλαξη των θαλασσίων συνόρων της στο ελληνικό πολεμικό ναυτικό και στο λιμενικό σώμα επιπλέον η ελλάδα να αξιοποιήσει τη ρήτρα παρέκκλησης του άρθρου 72 της συνθήκης και να σταματήσει να εφαρμόζει το δουβλίνο 3 για λόγους δημοσίας τάξεως και εσωτερικής ασφάλειας. ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ακολουθεί η κυρία Μπιλμπάου Μπαραντίνικα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το κόμμα μου ήδη από την δεκαετία του 1930 υποστηρίζει το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Αλλά εμεί θέλουμε να εκφράσουμε την ανησυχία μας για μια απόφαση η οποία αποδυναμώνει την ε, ευρωπαϊκή πορεία και την ε, ισότητα των πολιτών. Το Κοινοβούλιο έχει βέβαια τη δυνατότητα να βελτιώσει ένα κείμενο το οποίο ενεγράφει περισσότερο για να αντιμετωπίσει περισσότερα εσωτερικά προβλήματα του Κάμερο στον Ηνωμένο Βασίλειο από ότι των Ευρωπαίων. Για μια ακόμα φορά η Βρυξέλλες χρησιμοποιήθηκε σε μια εθνική συζήτηση ως ε, αποδιοπομπαίος τράγος για προβλήματα τα οποία έχουν προκύψει στην ίδια τη Μεγάλη Βρετανία. Το ευρωπαϊκό όραμα το οποίο υποστηρίζουν πολλοί λαοί χωρίς κράτος τονίζει ότι δεν θα πρέπει να γίνει δεκτή αυτή η αντιμετώπιση των Βρετανών. Θα πρέπει να ανοίξει όμως και η συζήτηση για τους λαούς χωρίς κράτη στην Ευρώπη που θέλουν να δεχτούν την ευρωπαϊκή ιδέα. Οι Καταλανοί, οι, οι Ουαλοί και οι Σκοτσέζοι και αυτοί έχουν το δικαίωμα να εκφράσουν ελεύθερα τη γνώμη τους για αυτά. Η κυρία Γκονσάλες Πένιας για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι αυτό το Σαββατοκύριακο καταλήξαμε σε μια συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο που λέει πολλά για το είδος Ευρώπης που κατασκευάζεται. Είναι η Ευρώπη των δύο ταχύτητων που μιλήσαμε για αυτή τη ταχύτητα της κρίσης να πραγματοποιήθηκε. Το περιθώριο ελιγμών των χωρών του, του Νότου έχει περιοριστεί ιδιαίτερα με απειλές και με ε, επιβολές. Η συνθήκες που δέχτηκε το Συμβούλιο αυξάνουν την ανισότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μονάχα για το εισόδημα των πολιτών αλλά και για το καθεστώς των πολιτών. Υπάρχουν 180.000 πολίτες από την Ισπανία ήδη στο Ηνωμένο Βασίλειο οι οποίοι θα γίνουν πολίτες της Ευρώπης δεύτερης κατηγορίας ενώ είναι άτομα τα οποία εργάζονται και βοηθούν την ευμάρεια του Ηνωμένου Βασιλείου. Δεν μπορούμε παρά να καταγγείλουμε την ε, ε, αυθαιρεσία αυτής της απόφασης που στρέφεται κατά του άρθρου 45 48 της Ευρωπαϊκή Συνθήκης. Δεν, αυτό επιβάλλει ακόμα μεγαλύτερα βάρη για τι χώρες της λιτότητα, χωρί κανένα αντιστάθμισμα. Ακολουθεί ο κ. Μπάλτσο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Θα ήθελα να αναφερθώ στο έγγραφο το οποίο έγινε δεκτό στη συνάντηση κορυφής. Οι σχέσεις ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να σέβονται ε, την κυριαρχία των κρατών μελών. Για το Ηνωμένο Βασίλειο αυτό σημαίνει ότι δεν θα συμμετέχει στις προσπάθειες περαιτέρω ολοκλήρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό δυστυχώς όμως δεν θα μπει στις συνθήκες ε, όταν αναθεωρηθούν την επόμενη φορά. Το θέμα λοιπόν δεν είναι συμβολικό απλά Είναι όμως σημαντικό ότι οι νόμοι οι οποίοι οδηγούν σε μια πιο εμβαθυμένη Ευρώπη δεν θα ισχύσουν για το Ηνωμένο Βασίλειο. Από την άλλη πρέπει να πούμε ότι αυτό θα δημιουργήσει διακρίσεις εις βάρος των χωρών οι οποίες έχουν ε, συμφέροντα αντίστοιχα με αυτά των Βρετανών. Er, er Εφόσον είναι ο κύριος Τσάβας εδώ, Κοιτάξτε, είναι προφανές ότι τα πράγματα εξελίσσονται με αντίθετο τρόπο αυτό που αναμενόταν η συμφωνία της διασκέψης κορυφής δεν καθησυχάζει τις ανησυχίες. Βεβαίως οι παραχωρήσεις θα επιβαρύνουν κυρίως τις νέες χώρες μέλη. και καλύτερα θα είναι η, Ευρωπαϊκή, η, ε, η Μεγάλη Βρετανία εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές προκλήσεις του παγκοσμιοποιημένου κόσμου. Ωστόσο, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, διότι η συμφωνία αυτή δεν πρέπει να ανοίξει την πόρτα για ειδικέ απαιτήσει άλλων χωρών μελών, οι οποίε να ικανοποιηθούν επίση. Σα. ευχαριστώ πολύ, η Προεδρεύουσα, ο κύριος Λόπες Αγγιλάρ, για ένα λεπτό. Νομίζω ότι είναι μια σημαντική ευκαιρία αυτό το οποίο συνέβη. Ε, δεν είναι η καλύτερη συμφωνία, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι προτιμότερο από την πιθανή έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου. Το θέμα είναι λοιπόν ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα που αντιμετώπισε ο κύριος Κάμερον και στην Κάτω Βουλή αλλά κυρίως στο εσωτερικό του δικού του πολιτικού κόμματος. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σέβεται το ευρωπαϊκό δίκαιο και στα πλαίσια της εφαρμογής των συμπερασμάτων ε, των αποφάσεων αυτών, να μην παραβιάζεται ε, η βασική αρχή της ελεύθερης διακίνησης και να μην μετατρέπονται οι μετανάστες να μην δίδονται στους μετανάστες και στους ίδιους Ευρωπαίους πολίτες λιγότερα δικαιώματα από ό,τι στους Βρετανούς πολίτες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και δυστυχώς και τα θέματα της κρίσης της μεταναστευτικής δεν έχει υπάρξει λύση λόγω του μη σεβασμού των ηλυμένων αποφάσεων. λεπτό. Ευχαριστώ. Η δήλωση που ακολούθησε τις διαπραγματεύσεις είναι ότι και οι δύο πλευρές ήταν ικανοποιημένες με τη συμφωνία. Αλλά οι αντιδράσεις των Βρετανών πολιτών μας δείχνουν ότι υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός Βρετανών που δεν είναι ικανοποιημένοι με αυτή τη συμφωνία. Ακόμα και αν μείνει το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να μεταρρυθμίσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το φεδεραλιστικό μοντέλο που πολλοί από τους ε, ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζήτησαν και πολλοί βουλευτές είναι επεπαλαιωμένο, δεν είναι προσαρμοσμένο στις σύγχρονες εποχές. Θέλουμε μεγαλύτερη αποκέντρωση της πολιτικής εξουσίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ας μην αυταπατώμετα. Αν το Ηνωμένο Βασίλειο μείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό δεν σημαίνει ότι τα εκατομμύρια Βρετανών που επικρίνουν την τωρινή κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα σιωπήσουν. Αλλά και αν το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσουμε να ζητούμε μεταρρυθμίσει οι υπόλοιποι. Ο κύριος Χουντής. Χωρίς μικρόφωνο. Χωρίς μικρόφωνο ο κύριος Χουντής. Είναι υποκριτική, ήταν και είναι υποκριτική στο προσφυγικό, το ξέραμε. Τώρα με την απόφαση την τελευταία, με τις δικές σας δηλώσεις, θέλετε να μας πείτε ότι είσαστε αδύναμοι ή και ανίκανοι να εφαρμόσετε μια ευρωπαϊκή λύση για το προσφυγικό. Πού είναι οι πανίσχυροι, άτεκτοι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιβάλλετε μνημόνια, που επιβαλλεται μνημονια εκβιαστικά πολιτικές λιτότητας. Τώρα φταίνε άλλοι ή τώρα εσείς δεν μπορείτε να το κάνετε. Οι δικές σας ευθύνες. Στην Ελλάδα το Γενάρη ήρθαν 68.000 πρόσφυγες. Έχουν εγκλωβιστεί στα σύνορα 6.000 και προβλέπετε με αυτή την πολιτική να εγκλωβιστούν ένα εκατομμύριο. Και εσείς τι κάνετε προκλητικά, θέλετε να επαναφέρετε σε λειτουργία τον κανονισμό του Δουβλίνου. Τι άλλο κάνατε, εμπλέξατε δυστυχώς με τη σύμφωνη γνώμη και της ελληνικής κυβέρνησης το ΝΑΤΟ, στρατιωτικοποιώντας το Αιγαίο, οξύνοντας το προσφυγικό πρόβλημα εκ των πραγμάτων και βάζοντας την ευρώπη και τη χώρα μου σε γεωπολιτικές ανακατατάξεις. πείτε καθαρά λοιπόν ότι με αυτά που κάνετε θέλετε να φορτώσετε όλο το βάρος στην ελλάδα σε ποια ευρώπη οδηγείτε τα πράγματα. ευχαριστώ πολύ. Ακολουθεί ο κύριος Κωνσταντίνος Παπαδάκης για ένα λεπτό. αποφάσεων του συμβουλίου και όχι η παραβίασή τους που έχει οδηγήσει στο μαζικό εγκλωβισμό χιλιάδων απελπισμένων προσφύγων στην ελλάδα. το συμβούλιο ενέκρινε τις συστάσεις της 12 ης Φλεβάρη που εφαρμόζοντας τη σέγγεν προβλέπουν συνοριακούς ελέγχους δίνοντας πράσινο φως για όλα κλειστά σύνορα φράχτες πλαφών προσφύγων ξεδιάλεγμα όσων έχουν τις προδιαγραφές φθηνού εργατικού δυναμικού για τα μονοπόλια με κατάσχεση των όποιων υπαρχόντων τους και απελάσεις των υπολείπων αυτή είναι η καπιταλιστική βαρβαρότητα που φέρνει τον υπεριαλιστικό πόλεμο την αιτία της προσφυγιάς και από πάνω με τη συμφωνία και της ελληνικής κυβέρνησης ο λύκος νάτο στο αιγαίο να αφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα της ελλάδας ενθαρρύνοντας την προκλητικότητα της τουρκίας αυτή είναι η ευρωπαϊκή ένωση και το νατο. στα δεσμά τους οι λαοί βρίσκονται σε διαρκή κίνδυνο. συνεπώς απαιτείται διαρκής λαϊκή πάλη κατά των υπεριαλιστικών πολέμων στήριξη των ξεριζωμένων σε αντιπαράθεση με τις ρατσιστικές φασιστικές δυνάμεις και διεκδίκηση μέτρων για απευθεία μεταφορά των προσφύγων στα κράτη τελικού προορισμού του κύριε κυρία για Πρόεδρε, Αντιπρόεδρε Ντομπρόφσκης, η κοινή δράση οφείλει να είναι ο οδηγός μας. Όμως όσα συμβαίνουν, μόνο την κοινή δράση δεν αναδεικνύουν. Τι θα γίνει με την υποχρεωτική μετεγκατάσταση στο προσφυγικό, είναι έτοιμη η κομισιόν να ενεργοποιήσει μηχανισμό κυρώσεων δηλαδή περικοπή κονδυλίων από τις αγροτικές επιδοτήσεις και τα διαρθρωτικά ταμεία για τα κράτη μέλη που αρνούνται να πάρουν πρόσφυγες στο έδαφος τους ή δημιουργούν εμπόδια όπως είναι το δημοψήφισμα στην ουγγαρία. τι θα γίνει με τη φρούρηση των συνόρων; μπορεί το νάτο να αναλάβει δράση με βάση τα συμφωνηθέντα ξεπερνώντας τις εκτός διεθνούς νομιμότητας αντιρρήσει που εγείρει η τουρκία; ένα πρέπει να είναι το μήνυμά μας δεν χωρούν παλινδρομήσεις από τα αρχικό συμφωνηθέντα στο νατο ούτε κολλησιεργίες από τα κράτη μέλη. σας ευχαριστώ. Μπρένερ, ένα λεπτό. Δεν είμαι μόνος εγώ που ανησυχώ για την κατάσταση στην οποία έχει περιπέσει το κόμμα της Ένωσης στη Βόρεια Ιρλανδία. Είναι εναντίον της παραμονής της Μεγάλης Βρετανίας. Παρ' όλα αυτά λέγεται ενωτικό κόμμα. Αν φύγει λοιπόν το Ηνωμένο Βασίλειο αυτό θα οδηγήσει σε μια περαιτέρω δημιουργία δημοψηφίσματος και ε, στην Βόρεια Ιρλανδία και στη Σκοτία και αλλού Φυσικά αν φύγει η Σκοτία, αν δεν υπάρχει η σημαία του Αγίου Ανδρέα, δεν μπορεί να υπάρξει Ηνωμένο Βασίλειο. Πώς μπορεί λοιπόν ένα κόμμα όπως αυτό το ενωτικό ε, Ιρλανδικό κόμμα να πιστεύει ότι δεν πρέπει να υπάρχει ένωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Μορβάη. Είναι διαδικαστικό αυτό. Κοιτάξτε, εγώ υπέγραψα για το Catch the Eye, ζήτησα να μιλήσω στην αρχή του απογεύματο. Και ήταν, ποια ήταν η αρχή των επιλογής που επελέγει. Τι θα συμβεί σε αυτή την αίθουσα μετά, αν μία φορά πάνω από 50 από τους 750 κάτι ε, εμφανιστούν. Αν δεν υπάρχει δυνατότητα να μιλήσουν οι περίπου δύο ντουζίνες από εμά που εμφανιζόμαστε στην αίθουσα. Ευχαριστώ. Κυρία Μόρβαη, στη διαδικασία Catch the Eye ε, προσπαθούμε να ακουστούν όσο το δυνατόν περισσότεροι. Αλλά πρέπει να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε μια ισορροπία μεταξύ των μεγαλύτερων και των μικροτέρων ομάδων. Οι μεγάλες ομάδες είχαν τρεις ομιλητές, οι μικρότερες δύο ομιλητές. Από εκείνους που δεν ανήκουν σε καμία ομάδα, όπως συνάδελφος από την Ουγγαρία, από το ίδιο κόμμα και εσείς, ακούστηκε, και κάποιος άλλος από τους ε, μη ε, γεγραμμένους, τους ανεξαρτήτους μίλησε. Είσαστε το τρίτο άτομο από τα μέλη, τα ανεξάρτητα που ε, ακούστηκαν στη διαδικασία Eye. Νομίζω ότι ήταν δίκαιη η όλη κατανομή που ακολουθήθηκε στην Ολομέλεια. Επίτροπε κύριε Ντομπρόφσκης, έχετε το λόγο ούτως ώστε να ολοκληρώσετε την όλη συζήτηση εκ μέσω Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου. Όσον αφορά τι διαπραγματεύσει από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων συμφώνησαν, κατέληξαν μια συμφωνία για να ικανοποιήσουν τι ανησυχίε του Πρωθυπουργού του κ. Κάμερον και η απόφαση τώρα είναι στα χέρια του Βρετανικού λαού όπως υπόθηκε και από τον πρόεδρο τον κύριο Γιούνκερ. Αν το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος είναι θετικό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αμέσως θα υποβάλει νομοθετικές προτάσεις στο Ευρωκοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, ούτως ώστε να υλοποιηθεί συμφωνία. Όσον αφορά την κρίση των προσφύγων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή νυχθημερών εργάζεται για την αντιμετώπιση της κρίσεως και να αντιμετωπιστεί η ροή των προσφύγων και πιστεύουμε ότι η λύση μπορεί να είναι μόνο μια ευρωπαϊκή λύση. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να συνεργαστούν μεταξύ τους και να εφαρμόσουν τις ήδη ε, συμφωνηθήσεις λύσεις. Μπορούμε να βρούμε τα πρώτα θετικά σημάδια. Έχουμε καλύτερη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων. Έχουμε πολιτική επιστροφή. Έχουμε τα κέντρα διαλογή και καταχώρηση, τα hot spots και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει ε, προτάσεις πολύ σύντομα για την έτη περαιτέρω βελτίωση καταστάσεω. Θέλουμε να συνεργαστούμε και με τους εξωτερικούς εταίρους. Είναι υψίστη σημασία αυτό και η συνάντηση με την Τουρκία και τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως την 7η Μαρτίου θα είναι πολύ σημαντικό γεγονός σχετικά με αυτό. Θα πρέπει να δώσουμε μια συντονισμένη απάντηση στην, στο πρόβλημα που προκύπτει από την προσφυγική κρίση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Επίτροπε Ντομπόφσκης. Η συζήτηση έχει λήξει.